Καλημέρα συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Η ημερήσια διάταξή μας είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη σήμερα. Άρχεται η συνεδρίαση. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, ε, θεωρώ ότι η προκεινόμενη ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Έχω κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τη Δευτέρα το βράδυ έλαβε χώρα η πέμπτη και τελευταία τριμερής ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ε, μετά από κάποιες τελευταίες προσαρμογές, οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μία πρόσκαιρη συμφωνία, η οποία επιβεβαιώθηκε χθες από την Κορεπέρα. Το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης της πρώτης ανάγνωσης θα υποβληθεί εις την ψηφοφορία, κοινή ψηφοφορία Αφετ Budget, τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ, στο Στρασβούργο στην ΒΙΚ 200 ε, ε, και σε περίπτωση επιτυχούς ε, θετικής ψηφοφορίας, αν εγκριθεί δηλαδή από αυτήν την κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΑΦΕΤ Μπούτζ, τότε θα υποβληθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια πριν το τέλος της ιδίας συνόδου. Εδώ έχουμε τη συνάδελφο η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στους τριμερείς ε, διαλόγους που δεν είναι και εύκολο πράγμα γιατί αφορούσαν τρεις ε, επιτροπές και επομένως χρειάστηκαν τα ηγετικά της διαφυσβήτητα προσόντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί νομίζω ότι το καλύτερο νέο είναι ακριβώς ότι έχουμε συμφωνία και ότι επιτέλους χθε ε, έδωσε πράσινο φως ε, η, κορεπέρα. Πέντε τριμερείς ε, διάλογος, πολλές ενδιάμεσες συζητήσεις, 60 ώρες διαπραγμάτευσης. πολύ ε, σημαντικές γιατί έπρεπε να συμφωνήσουν τρεις εισηγητές από τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες με παρελθόν και background διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει ιδιαίτερα περίπλοκο ήταν το θεματικό. οι τεχνικές ε, ε, ομάδες βεβαίως έπαιξαν θεμελιώδη ουσιώδη ρόλο διότι οι πολιτικοί τριμερείς διάλογοι έβαζαν κάποιες θέσεις αλλά οι τριμερείς τεχνικοί διάλογοι γραμμή υπό γραμμή λέξη προς λέξη προσπάθησαν να βρουν την σωστή ε, διατύπωση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως ε, την ε, ομάδα μας του προϋπολογισμού. Βέβαια ρόλο έπαιξαν και οι τεχνικές ομάδες των άλλων δύο επιτροπών, αλλά εδώ είμαστε στη δικιά μας των προϋπολογισμών και γι' αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερως. Δύο μικρά σχόλια όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνία, διότι ε, ε, από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο δεν είχε μία ιδιαίτερα σημαντική κεντρική ε, ιδέα στην ουσία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις δεν είχαμε την δυνατότητα να ε, ε, ολοκληρώσουμε την διαπραγμάτευση. Ε, στο τέλος, στο τέλος θέσαμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας και επομένως πετύχαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Στην ουσία δηλαδή καταφέραμε να μετριάσουμε κατά πολύ αλλά και να εστιάσουμε περισσότερο τους ουσιώδεις στόχους και καταφέραμε επίσης να πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε επενδύσεις οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν την ανάπτυξη σε χώρες αποδοχής. Επίσης καταφέραμε να βελτιώσουμε πολύ τα κριτήρια της ε, λεγόμενης ε, κοινωνικής ε, ευθύνης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή για τα εργασιακά δικαιώματα, πράγματα δηλαδή που μπορεί να φαίνονται προφανή αλλά που εμείς θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί η συμπληρωματικότητα και η προσθετικότητα γιατί θα είναι πολλά τα ταμεία τα οποία θα συμπεριληφθούν επίσης ε, από το 20 πέρασε το Συμβούλιο στο 28% όσον αφορά ε, τα συστατικά των ε, επιχειρήσεων για την κλιματική αλλαγή. Επίσης συμφωνήσαμε με οτιδήποτε αφορά την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής μέσω θέσπισης συγκεκριμένων κανόνων και ε, ε, αντικειμενικών στόχων. Επίσης υπάρχουν και, υπάρχει και το, εσωτερικό ας πούμε, τμήμα, δηλαδή το γεγονός ότι στη Στρατηγική Επιτροπή θα έχει παρατηρηθεί το Κοινοβούλιο και επίσης ε, βάλαμε και θέσαμε και πάρα πολλές προϋποθέσεις ε, αξιολόγησης ε, στην Κομισιόν, πολλά προαπαιτούμενα δηλαδή αξιολόγησης έτσι ώστε να ξέρουμε, να έχουμε ένα λόγο όσον αφορά τα όσα θα λάβουν χώρα για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι στόχοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτά που μας είπατε, αλλά και για την ε, δέσμευσή σας, τη στράτευσή σας. Να σας πω επίσης ότι η αποστολή στο Ισραήλ του Ιουλίου, Ισραήλ και Παλαιστίνη, ε, μεταφέρεται, ε, αναβάλλεται, γιατί θέλουμε να πάμε και στη Γάζα και στην Υπεριορδανία και... Ε, θεωρήθηκε αδύνατη η προστασία της αντιπροσωπείας στην Γάζα ε, λόγω της παρούσης καταστάσεως και της, ε, των προβλημάτων στην ηλεκτρική τροφοδοσία στην Γάζα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι παρά να περιοριστούμε σε μια μικρή επίσκεψη η οποία θα ήταν συμπιεσμένη ας πούμε και θα αφορούσε μόνο την Περιοδάνεια καλύτερα θα ήταν να γίνει η αποστολή αυτή στην αρχή του 2018. Επίσης οι συντονιστές ε, αποφάσισαν, πήραν κάποιες αποφάσεις ε, για το ε, σώμα αλληλεγγύης θα είναι υπεύθυνη κυρία Βαϊτερή, για τα, τα συστήματα προμήθειας το, του Σώματος Αλληλεγγύης Λαβία Financial Budgetary Measures ε, όσον αφορά ε, τις, ε, τις προ, υφιστάμενες προκλήσεις ο άλλος η ομάδα S&D θα δώσει κάποιον υποψήφιο. Καθορισμός προγραμμάτων αναπτυξιακών όσον αφορά την ικανότητα αντίδρασης και άμυνας. Το ΕΛΚ θα είναι υπεύθυνο να ορίσει εισηγητή. Επίσης το ΕΛΚ θα προτείνει εισηγητή και για μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία ε, European Defense Action Plan. Ετήσια έκθεση για την ε, υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας, ο υποφαινόμενο ο πρόεδρός σα. υποψήφιο. Οι συντονιστέ. Ε, Επίσης έλαβαν κοινοποίηση ε, για την ε, η πρόσληψη ενός ε, ειδικού συμβούλου στην ιατρική υπηρεσία. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να μην, συζητηθεί, να μην ζητηθεί επιπλέον κονδύλιο. Επίσης για τη διαχείριση και έλεγχο των καταπιστευμάτων ε, ε, ζητήθηκε παρακολούθηση. Αυτό, παρακολούθηση. Αυτό θα γίνει ε, από την επόμενη χρονιά και μετά. Αυτές είναι οι αποφάσεις τις οποίες ήθελα να σας γνωστοποιήσω. Φτάνουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ πολύ να κάνουμε ένα μία προσπάθεια να δούμε αν είναι όλοι αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ε, 27 είναι οι κάρτες. 20... Α, εγώ δεν είχα βάλει την κάρτα μου, ορίστε. Πρώτο κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε.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 εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 88 υπέρ κατά α, α, δεν γίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 160 158 συγγνώμη απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 164 με μια προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 167 καταπίπτει. Συμβιβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές Α, ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη. Συμβιβαστική 19α. Υπέρ. Κατά. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της ε, συμβιβαστικής 19α. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ με μια προφορική τροπολογία υπέρ επί της διαδικασίας εμείς έχουμε υποβάλει τη 202, η οποία έχει ε, προσθε... στην οποία έχει προσθεθεί η προφορική τροπολογία, δηλαδή να ψηφίσουμε πρώτα μέχρι το outside EU budget και μετά το δεύτερο τμήμα χωριστά. Ποια είναι η άποψη του εισηγητού επί του θέματος αυτού. Συγγνώμη, για την 212 μιλάμε. Ναι. Και όπου υποτίθεται ότι υπήρχε προφορική τροπολογία του εισηγητή και μαζί με αυτήν θα μπορούσαμε να υπερψηφίσουμε την παράγραφο. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε τώρα να δεχτούμε χωρί τη ψηφοφορία να αποσυρθεί η προφορική τροπολογία. Τι ακριβώς ζητάτε για να το ξεκαθαρίσουμε. Κοιτάξτε, έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να γίνει χωριστή ψηφοφορία, κατά τμήματα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ζητούμε να ψηφιστεί η αρχική τροπολογία πρώτα και μετά η τροπολογία με την προστίκη. Πρόεδρος, εάν έχετε συμφωνήσει με τον εισηγητή, έτσι ώστε να εντάξει την προσθήκη ε, μπορεί να γίνει και αυτό και να κάνουμε δηλαδή μία και μόνη ψηφοφορία. Ενιαία ψηφοφορία όχι. Μία, μία, ψηφο, μία ψηφοφορία όχι δεν θέλουμε. Εμείς ζητούμε να ψηφιστεί η τροπολογία όπως ήταν αρχικά. Δηλαδή εμείς απορρίπτουμε την προφορική τροπολογία. Εάν, θέλει κάποιος να ψηφιστεί η προφορική τροπολογία να γίνει χωριστά. Κύριε Σιγητά. Λοιπόν, Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Εάν η Γκουε θέλει να αποσυρθεί η προφορική τροπολογία, ε, εντάξει, αν θέλετε να διατηρηθεί η προφορική τροπολογία, τότε εγώ θα ζητήσω υπερψήφιση. Αν θέλετε να αποσυρθεί η προφορική τροπολογία, που είναι το μόνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε τώρα, να αποσύρετε την προφορική τροπολογία, τότε εγώ θα δώσω αρνητική γνωμοδότηση. Donc, vous... Eh, Pedimos que se retire la, o sea, la, la enmienda del reporter y se vote la original. Sí. Εμείς θέλουμε να αποσυρθεί η, η προφορική τροπολογία και να ψηφιστεί η αρχική τροπολογία. Πρόεδρος, επομένως, ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία, δηλαδή την τροπολογία της κυρίας Ριάντα, επί, του οποίου γνωμοδότη, επί της οποίας τροπολογία είναι αρνητική η γνωμοδότηση. Ψηφίζουμε για την τροπολογία της κυρίας Ριάντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 213 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 214 υπέρ, κατά, θα θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 2.14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη 18 ψήφοι κατά, έναντι 8 ψήφων υπέρ. Τροπολογία 215 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 216 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 218 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία συμβιβασμός 26 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται τροπολογία 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις, παράγραφος 15 της ε, Επιτροπής Απασχόλησης, τροπολογία 15, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1 της γνωμοδότησης ε, ΦΑΜ, της Επιτροπής Γυναικών, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε επί του συνόλου του τροποποιημένου κειμένου. Ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία νομίζω λέει ο πρόεδρος. Ε. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν επί του συνόλου του κειμένου. Ψήφισαν όλοι. Όχι, ναι. Ωραία. Πέρασε της ψηφοφορίας. 22 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 2 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Θα ψηφίσουμε τώρα επί της τη της κυρίας Μόνικα Βάνα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή. τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επί του συνόλου του κειμένου άρχεται η ψηφοφορία διηλεκτρονικής ψηφοφορίας Εγκρίθηκε 24 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Βάνα. Φτάνουμε τώρα ε, στην έκθεση του κυρίου Γένσε Γκέγερ. Έχουμε τέσσερις μεταφορές. Ε, η μία φορά την Τουρκία. Η κυρία Τερέζα Μπάλ Ευχαριστώ πολύ. Πολύ γρήγορα κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, οι 7 και οι 11 ε, μεταφορές ε, αφορούν την διευκόλυνση για την Τουρκία. Για την 7 ήδη συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και αποφασίσαμε να την μεταθέσουμε. Εν πάση περιπτώσει, τελικά αποφασίσαμε να ψηφιστεί ε, και θέλουμε να υπερψηφιστούν οι δύο μεταφορές. Ένα σχόλιο μονάχα ήθελα να κάνω, γιατί καμιά φορά ε, διαβάζουμε μεταφορές και τέτοια ε, και δεν κατανοούμε ότι το Συμβούλιο αποφασίζει ε, να μην να μην ε, επιβάλλει, ε, να μην επιβάλλει τόκους ε, καθυστέρησης υπερημερίας στην περίπτωση της διευκόλυνσης για την Τουρκία ή διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε. Εμείς εδώ σπάμε τα, κεφάλια μας, προσπαθούμε να βρούμε χρήματα Και, τα και το Συμβούλιο σιγά σιγά και χαλαρά και όποτε θέλει και ε, στην ουσία ε, δεν επιβάλλει καμία, ε, καμία ποινή ας πούμε επί παραβάση ή οτιδήποτε. Με αυτό εμείς δεν συμφωνούμε. Εν πάση περιπτώσει με τις άλλες μεταφορές δεν έχουμε πρόβλημα. Η 8 την συζητήσαμε και μόλις εγκρίναμε κείμενο. Ε, και έχουμε και άλλη μία μεταφορά για την ε, βελτίωση των ε, στοιχείων IT και τα λοιπά. Νομίζω ότι μπορούμε να υπερψηφίσουμε και τις τέσσερις μεταφορές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν μεταφορά 7 του 2017 άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε 21 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Μεταφορά 8 του 2017 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ 3 κατά. Μεταφορά 10 του 2017, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 24 υπέρ 1 κατά εγκρίνεται. Μεταφορά 11 του 2017 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρασε. 23 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά εγκρίνεται. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ίντρεκ Τάραντ για τις ε, μεταφορές ε, άλλων τμήματων. Στην τελευταία συνεδρίαση της ε, η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Δημοσιονομικού Κανονισμού ε, έχει ε, αναφέρει προβλήματα σε, τρία, ε, σε τρεις αιτήσει χρηματοδότησης βάση του άρθρου 27. Κύριε Τέρεντ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι όπως το βλέπω εγώ μπορούμε όλοι να ψηφίσουμε, να υποστηρίξουμε τη μεταφορά υπαρθμών 3 και δεν θα βγάλω ομιλία, απλά σας ε, ζητάω να καταψηφίσετε το 1 και 2 γιατί η Επιτροπή των Περιφερειών εδώ έχει δώσει εξηγήσει ε, που δεν είναι ικανοποιητικέ. Καθώς οι αρχές του προϋπολογισμού είχαν καθορίσει ε, συγκεκριμένους πόρους για αυτές τις ε, δραστηριότητες και δεν πρέπει να ζητάνε περισσότερα. Αυτά είναι ολίγης. Αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα, μπορώ να σας πω ότι κόβουν προγράμματα για μαθητές για να δημιουργήσουν ε, γραφικά, γραφιστικά για πολιτικές ομάδες. Εντάξει, και εμένα μου αρέσουν οι συνάδελφοι εδώ πέρα, αλλά δεν χρειάζεται να βελτιωθεί η οπτική του ταυτότητα όπως τη λένε. Ο κύριος Ντεπρέ. Κύριε Πρόεδρε δεν θα αναφερθώ, δεν θα εκφράσω άποψη εις, ε, όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά επί της αρχής. Ε, γιατί εδώ παίζεται μία αρχή. Εμείς έχουμε ένα ε, άρθρο του προϋπολογισμού, βάσει του οποίου εμείς δώσαμε, εγκρίναμε ένα, μια πίστοση, ένα κονδύλι, η οποία 500.000 ε, ευρώ νομίζω είχαν ζητηθεί και εμείς ε, ε, είπαμε 300.000 ευρώ. Το εγκρίναμε και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Τι κάνει λοιπόν η, το, το Συμβούλιο των, Επιτροπή των Περιφερειών για να μπορέσει να, να βρει αυτό το αρχικό κονδύλι το οποίο εμείς περικόψαμε και δεν εγκρίναμε προσπαθεί να βρει χρήματα από άλλα κονδύλια. Τη στιγμή λοιπόν που εμείς αποφασίσαμε ότι ότι το αρχικό αίτημα ε, δεν ήταν σωστό και έπρεπε το ποσό να μειωθεί ε, ε, και ε, προσπαθούν να βρουν άλλες μεταφορές έτσι ώστε να φτάσουν στο αρχικά ετηθέν ποσό υπάρχει ένα πρόβλημα επί της αρχής και αυτό με ενοχλεί. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά λέω ότι ανεξάρτητα από την ουσία και από το αίτημα το συγκεκριμένο εγώ έχω την τάση να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Τάραντ. Ζητά κάποιος άλλος το λόγο, ο κύριος Τάραντ τελευταία παρατήρηση. Συμφωνώ με τον κύριο Ντιπρέ και για να σας αποδείξω αυτό το οποίο έλεγα, ο κύριος Κρόνσπερξ Έλμας ε, μου είπε ότι παρά την απόφασή σας ήδη δαπανούμε τα λεφτά. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχει ζητηθεί ε, ε, ονομαστική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως. επιμένετε σε αυτό, το επιβεβαιώνετε. Roll call vote λοιπόν. Η πράσινη, η γκούε, ε, η ECR έχει ζητήσει ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως. Επί της πρώτης μεταφοράς λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 15 ψήφοι υπέρ, 9 κατά 2 αποχές. Δεύτερη μεταφορά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 ε, ψήφοι υπέρ, 6 ε, ψήφοι κατά 2 αποχές εγκρίνεται. Τρίτη. Άρχεται. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Η κυρία Χολμάγερ είναι εδώ. Madame n'a pas pu nous Όχι. Προτείνει πάντως η κυρία Χολμάγερ να μετατεθούν οι αποφάσεις μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, διότι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ερευνητική της εργασία. Ε, συμφωνείτε, συμφωνούν τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών να μεταφερθεί η ψηφοφορία επί των δύο ε, κονδυλίων. Δέχεστε. Δέχεστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν ε, με την διαδικασία της ψηφοφορίας και τώρα θα συζητήσουμε για μία μελέτη την οποία είχαμε ζητήσει σχετικά με τις συνέργειες ανάμεσα στους στόχους που τέθηκαν στην ετήσια επισκόψη ανάπτυξης και τον συντονισμό ανάμεσα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Το 2016, στα πλαίσια της συζήτησης ε, ε, της εμπλοκής ε, της Επιτροπής των Προϋπολογισμών στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν μία μελέτη ακριβώς για τις συνέργειες που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στους στόχους της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και της συνεισφοράς των προϋπολογισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών στον εν λόγω, στην επισκόπηση. Ε, λοιπόν, θα γίνει μία παρουσίαση από τον δόκτωρα Χάφνερ, ο οποίος είναι lead ε, economic modeler στο ε, Cambridge, μετά ο Ματέο Μπαρμπέρι, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής της Ομάδας Ερευνών. Η Επιτροπή Οικονομικών, συγγνώμη, μετά από δικό μου αίτημα, η Κομισιόν ε, ε, ζήτησε από την Κομισιόν μάλλον ε, να ορίσει κάποιον εκπρόσωπο. Είναι ο κύριος Ζωάν Μπουρέλ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη Γενική Διεύθυνση Budge και θα έχουμε επίσης και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΦΙΝ. Η παρουσίαση της ε, μελέτης μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για να δούμε ποια μπορεί να είναι η συμβολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών ε, στην, ε, στο γενικότερο θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πράγμα που θα αποτελέσει αντικείμενο και τη επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Πραγματικά, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ αναρωτήθηκα εάν πραγματικά η έκθεση αυτή είναι απαραίτητη τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει και στους εθνικούς προϋπολογισμούς αλλά και στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαιτήσει θέμενη αξία δεν μου φάνηκαν να καλύπτονται σε αυτή την περίπτωση και ευελπιστώ ότι η μελέτη που θα μας παρουσιάσουν τώρα οι ε, μελετητές ελπίζω λέω, ευελπιστώ ότι θα απαντήσει ε, σε αυτά τα ερωτήματα. Ο κύριος Μάρκο Χάφνερ νομίζω είναι μαζί μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί η εν λόγω μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, ε, δηλαδή η ανάπτυξη και η σχέση με το ΑΕΠ είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα θέλαμε ε, στο μέλλον ε, να διατίθεται και online αυτή τέτοιου είδου έγγραφο, ώστε να μπορούμε να προετοιμαστούμε και προκειμένου να μπορούμε να ενημερώσουμε και του ευθύνοντε στις πατρίδες μας. Οπότε σας παρακαλώ στο μέλλον πάντοτε να, ε, να διατίθεται online. Votre souhait légitime est enregistré, Rubig. Monsieur le docteur Marco Hafner. Ο κύριος ε, Μάρκο Χάφνερ. Σας ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Χάφνερ, που είστε μαζί μας. Έχετε στη διάθεσή σας κάποια λεπτά, θα τα βρω, 20 λεπτά, έτσι ώστε να παρουσιάσετε την έκθεσή σας και το περιεχόμενό της. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνατε τη δυνατότητα σήμερα να παρουσιάσουμε τα πορίσματα της ε, μελέτης μας σε ό,τι αφορά τις ενέργειες ανάμεσα στους στόχους που αναφέρονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τον ε, προπολογισμό τόσο της Ένωσης όσο και τους εθνικούς προπολογισμούς. Okay. Sorry about this uh, problem with the, with the slides. So first of... Ζητώ συγγνώμη, είχα ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα εδώ με τις ε, διαφάνειες. Άρα, ε, ποια είναι η αναδομή της παρουσίασης. Καταρχήν θα αναφερθώ στο γενικότερο πλαίσιο της μελέτης. Ε, θα αναφέρω τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε για να διεξάγουμε την έρευνά μας. Θα αναφερθώ στα απορίσματα και ε, στις, ε, στο τι αυτό σημαίνει στο επίπεδο της πολιτικής και αν έχουμε αρκετό χρόνο θα εξετάσουμε και περαιτέρω ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το γενικό πλαίσιο καταρχήν αυτή τη μελέτη. Ε, να πούμε ότι ε, τη επισκόπηση τη ανάπτυξη αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και κατά συνέπεια ε, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία μέσω ακριβώς των παρεμβάσεων στον προπολογισμό ε, και τη εξήγησης του προπολογισμού. Και στο πλαίσιο αυτό ε, δίνει και καθοδήγηση στα κράτη-μέλη μέσω συστάσεων αναχώρα ε, προκειμένου να επιτύχουν θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα. Πέραν όμως τις Έμεση άσκηση πολιτική μέσω δηλαδή τη συμμόρφωση με το Σύμφωνο σταθερότητα ε, και ανάπτυξη ε, και τι περαιτέρω διαδικασίε κατά παρόβαση, τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλα περιθώρια ευελιξία σε ό,τι αφορά την πολιτική που εφαρμόζουν. Και το ίδιο ασχεί για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή παρότι αναφέρονται συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένε προτεραιότητε, αυτό δεν σημαίνει ότι απηχούνται σε κάθε περίπτωση στον, ε, είτε στον ετήσιο προπολογισμό είτε στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε εμεί θεωρήσαμε πως θα ήταν σημαντικό να δούμε κατά πόσο η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη απηχείται και οι συστάσει αναχώρα απηχούνται στου ε, προπολογισμού δηλαδή, τη Ένωση και των κρατών Άρα λοιπόν ε, ουσιαστικά οι στόχοι της ε, ε, έρευνάς μας ή της μελέτης μας διατυπώθηκαν ως τέσσερα ερωτήματα. Καταρχήν ήταν το ερώτημα του κατά πόσο ο προπολογισμό της Ένωσης απηχεί τους τομείς προτεραιότητας προκειμένου να δημιουργηθεί οικονομική ανάπτυξη και κατά πόσο από την άλλη πλευρά οι εθνικοί προπολογισμοί ανταποκρίνονται στα, στις αντίστοιχες συστάσεις χώρα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν κατά πόσο αυτοί οι προπολογισμοί ακολουθούν τις κατευθυντήρες γραμμές της Ετήσιας Επισκοπής της Ανάπτυξης ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία και ε, να υπάρχουν και κατάλληλε δεσμεύσει κονδυλίων στον προπολογισμό. Το τρίτο ερώτημα ήταν κατά πόσο υπάρχουν συνέργειε ανάμεσα στον προπολογισμό τη Ένωση και του εθνικού προπολογισμού, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι που αναφέρονται στην ετήσια επισκόπηση και στι συστάσει χώρα. Και τέταρτο ερώτημα, κατά πόσο τα μέτρα αυτά που υιοθετήθηκαν έχουν πραγματικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ή την πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ε, ποιότητα της ε, δημόσια δαπάνη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεθόδους της μελέτης. Γενικά λοιπόν ο στόχος μας ήταν να συλλέξουμε πληροφορίες από μια σειρά από διαφορετικές πηγές. Όπως για παράδειγμα είχαμε εδώ, εξετάσαμε μακροοικονομικά ε, μακροοικονομική τεκμηρίωση από την πλευρά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ε, εκθέσεις για τις ε, κάτω χώρες από την Επιτροπή και ούτω καθεξής. Επίσης είχαμε και δεδομένα της Eurostat σε ό,τι αφορά και πάλι δημοσιονομικά στοιχεία και προσπαθήσαμε να εξετάσουμε ποια ήταν τα στοιχεία που αναφέρονταν στις συστάσεις αναχώρα αλλά και τα στοιχεία που αναφέρονταν στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη για να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό λήφθηκαν υπόψη για την πρόθεση της ανάπτυξης. Και εδώ θα πρέπει να πούμε βλέπουμε ότι καλύψαμε στην ανάλυση μας την περίοδο 2014-2017 ε, και οι συστάσεις αναχώρα και η εφαρμογή του σε ό,τι αφορά το 2016 δεν είναι πλήρης ε, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί, είχαν ολοκληρωθεί ακριβώς τα προγράμματα που είχαν ξεκινήσει για το 2007 σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των προπολογισμών. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα το γεωγραφικό ε, πεδίο αν θέλετε, εφαρμογή τη μελέτη. Καλύψαμε το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από εκεί και μετά κάναμε και κάποιε πιο στοχευμένε ε, εξετάσεις αν θέλετε χωρών, δηλαδή 12 ε, μεγάλα κράτη-μέλη και 12 μικρά κράτη-μέλη λαμβάνοντας υπόψη και περαιτέρω παραμέτρους όπως τη γεωγραφική τους κατανομή. Ε, από εκεί και μετά θα πρέπει να πούμε ότι ε, ε δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στις τάσεις αναχώρα που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Για να σας ε, ε, αναφέρω ένα παράδειγμα, εάν έχουμε συστάσεις οι οποίες αναφέρονται για παράδειγμα στην περαιτέρω προώθηση των δράσεων για ε, έρευνα και ανάπτυξη, ναι, θα είχε συμπεριληφθεί, αλλά αν υπάρχει για παράδειγμα κάποια σύσταση σε ό,τι αφορά την βελτίωση τη ποιότητα τη ε, εκπαίδευση, δεν θα έχει ληφθεί υπόψη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα απορίσματα. διαπιστώσαμε ότι ο προπολογισμό τη Ένωση απηχεί τι ε, προτεραιότητε τη ε, επισκόπηση ανάπτυξη με διάφορου τρόπου. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά του τρει βασικού ε, τομεί, δηλαδή διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη, ναι, ανταποκρίνεται στα διάφορα καλέσματα για επενδύσει ο προπολογισμό. Δηλαδή, υπάρχουν μία σειρά από γραμμέ του προπολογισμού που μπορούν να θεωρηθούν σχετικέ, ειδικότερα τα 1α, 1β και 2 ε, που αναφέρονται ειδικότερα ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις ε, ή μάλλον στα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Από εκεί και μετά τα σχετικά κονδύλια αυξήθηκαν και σε απόλυτους αριθμούς και κάτι διάρκεια τη εκτέλεση του υπολογισμού. Δηλαδή, ε, κατά τα τρία ε, χρόνια που εξετάσαμε, η αύξηση των ε, δαπανών στι εν λόγω γραμμέ αυξήθηκε περισσότερο σε σύγκριση με το σύνολο του υπολογισμού. Αλλά από την άλλη πλευρά, η εν λόγω αύξηση είχε γίνει ήδη από την αρχή του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί δεν υπάρχουν μεγάλα περισσότερα ευελιξία σε ό,τι αφορά την αύξηση των σχετικών κοντιλίων αυτών των συγκεκριμένων γραμμών. Από εκεί και μετά ε, υπάρχουν και κάποιε θεσμικέ ε, συμφωνίε σε ό,τι αφορά την, ε, τον προπολογισμό τη Ένωση, ακριβώ επειδή συμφωνείτε και στο πλαίσιο του πολιετού ε, δημοσιονομικού πλαισίου, δεν είναι εύκολο να ληφθούν υπόψη ε, τάσει βραχυπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά όμω έχει εκφραστεί η βούληση να και υπάρχει πρόθεση να ε, προσαρμόζεται καλύτερο προπολογισμό στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη, θέτοντα για παράδειγμα κάποια όρια σε ό,τι αφορά όρια δαπανών σε ό,τι αφορά νέε πρωτοβουλίε όπω το Εράσμου ή το Ευρώπη 2020. Από εκεί και μετά η δημιουργία δύο νέων δημοσιονομικών εργαλείων Όπω η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τι Στρατηγικές επενδύσει αποτελούν τρόπου περαιτέρω κινητοποίηση των κονδυλίων προκειμένου ακριβώ να ανταποκριθεί ο προπολογισμό στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα εξετάσαμε το κατά πόσο οι προτεραιότητε τη ετήσια επισκόπηση απηχούνται στον προπολογισμό τη Ένωση. Η γενική λοιπόν απάντηση είναι ναι. Τώρα εξετάζουμε τι προτεραιότητε των εθνικών προπολογισμών και τη συμμόρφωσή του με τι συστάσει αναχώρα και την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη. Γενικά λοιπόν διαπιστώσαμε στη μελέτη μα ότι τα εφιστάμενα επίπεδα τη ε, ε, επίπεδα αν θέλετε της εφαρμογής ή της υλοποίησης των συστάσεων αναχώρα ε, δεν είναι πλήρως ικανοποιητικές. Δηλαδή αν δούμε τα σχέδια των προϋπολογισμών και τα, και τα συστήματα μεταρρύθμισης μόνο σε 21 από τα 106, ε, από τις 106 συστάσεις έχουν ξεκινήσει οι αντίστοιχες δράσεις. Ε, ενώ στα 3 ε, τέταρτα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση, δεν έχει, ή έχει σχεδιαστεί, ενώ σε 2 δεν έχει ξεκινήσει καν. Εδώ 4 CSR, συστάσεις, ούτε έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός τους, ούτε φυσικά και η υλοποίησή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τη επιτροπή σε ό,τι αφορά την πρόοδο των κρατών μελών σε σχέση με τις συστάσεις αναχώρα, μόνο τέσσερι συστάσει ε, ε, θεωρούνται, δηλαδή 4% θεωρούνται ότι δεν έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο, σε 52 υπήρξε αρκετή πρόοδο και σε 37 ε, περιορισμένη πρόοδο, ενώ σε 5 καμία πρόοδο. Από εκεί και μετά υπάρχουν λοιπόν κάποια κενά εδώ σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συστάσεων και όταν εξετάσουμε αυτές τις ε, τάσεις και σε, αυτό το, ε, σε ό,τι αφορά το περιορισμένο ε, δείγμα των 12 κρατών μελών, διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται περισσότερο με τις συστάσεις όταν βρίσκονται σε κάποια εξαιρετική διαδικασία, όπως για παράδειγμα τη διαδικασία του υπερβολικού έλλειμματος. τώρα, μετά από, την, ε, από αυτή την εξέταση που έγινε από την Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά την ε, συμμόρφωση των κρατών μελετών με συστάσει ένα χώρα, να πούμε ότι βρήκαμε κάποιε αποκλήσει. Δηλαδή, σε 47% των περιπτώσεων οι αξιολογήσει είχαν ολοκληρωθεί και ενώ η υλοποίηση 72 συστάσεων έχει ξεκινήσει στα κράτη-μέλη, μόνο σε 52 διαπίστωσε πραγματική πρόοδο η Επιτροπή. Ταυτόχρονα σε 37 συστάσεις αναχώρα η Επιτροπή διαπίστωσε περιορισμένη ε, πρόοδο σε αντίθεση με τα κράτη-μέλη που είχαν αναφέρει ένα υψηλότερο αριθμό. Άρα λοιπόν σε ε, γενικές γραμμές εξολογήσεις που γίνονταν και το, και το κείμενο της εξολόγησης από την πλευρά των κρατών μελών ήταν πιο θετικό από ό,τι εξολόγηση της Επιτροπής. άρα λοιπόν ο στόχος βέβαια εδώ είναι να, ε, μέσω και των δικτών να γίνεται η σχετική αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Αλλά ένας ακόμα τρόπος για να εξετάζεται η πρόοδος σε ό,τι αφορά δηλαδή την εφαρμογή των προτεραιοτήτων της ετήσιας επισκόπησης με πιο κενικό τρόπο είναι να εξετάζουμε τους δημοσιονομικού δείκτε, του δείκτε δηλαδή του προπολογισμού και την εξέλιξή του σε σύγκριση ή σε σχέση με αυτέ τι προτεραιότητε. Σε αυτή λοιπόν τη διαφάνεια βλέπετε ποιε ήταν οι ε, αλλαγέ που έγιναν εκεί σε αυτού του δείκτε ε, και τα χρώματα ανταποκρίνονται ακριβώ ε, σε αυτή την πρόοδο. Δηλαδή, όταν έχουμε κίτρινο κουτί σημαίνει ότι δεν υπήρξε πρόοδο, είναι η ίδια κατάσταση. Πράσινο κουτί σημαίνει ότι υπήρξε αύξηση, ενώ κόκκινο σημαίνει ότι υπήρξε μείωση των κονδυλίων. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε και πάλι ότι δεν υπάρχει ομοιόμορφη ε, λήψη υπόψη των προτεραιοτήτων της ετήσιας επισκόπησης στους εθνικούς προπολογισμούς. Από εκεί και μετά υπάρχουν κάποιες επιμέρους συστάσεις χώρα που έχουν εφαρμοστεί από, τις, ε, απο από διαφορετικά κράτη-μέλη. Ε, και εκεί δηλαδή όμως διαπιστώνουμε σε σχέση δηλαδή με την εφαρμογή των συστάσεων ε, μια διαφορετική εικόνα ανά κράτος μέλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν ε, συνέργειε ανάμεσα στον προπολογισμό τη Ένωση και του εθνικού προπολογισμού. Αλλά βέβαια ο προπολογισμό τη Ένωση περιμένει μικρό σε σύγκριση με του εθνικού προπολογισμού. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αναμένεται πω θα εστιάζει περισσότερο σε τομεί προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, σε περιπτώσει εκείνε, ε, δηλαδή έργων που ήδη χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη και τα οποία μπορούν να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων. Άρα λοιπόν ε, εάν ε, το δούμε πολύ ε, εξειδικευμένα, πολύ περιορισμένα, ναι υπάρχουν συνέργειες μεταξύ προϋπολογισμού Ένωσης και προϋπολογισμών κρατών μελών. Μέσω ακριβώς και της εφαρμογής των διαθροτικών και επενδυτικών ταμείων και μέσω της επιχειρησιακής εφαρμογής των εκτέλεσης των προϋπολογισμών στα κράτη-μέλη. Και ο προπολογισμό, ε, ε, το κατά πόσο ο ε, προπολογισμό τη Ένωση συμβάλλει ή υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην εκτέλεση των προτεραιοτήτων τη ετήσια επισκόπηση είναι δύσκολο να αξιολογηθεί. Ειδικότερα αφού έχουμε και τις διάφορες ερεσιμότητες που προβλέπονται. Και βέβαια τώρα το νέο εργαλείο, δηλαδή το Ταμείο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμα τρόπο αύξηση αυτών των συνεργειών, αλλά δεν μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί η χρησιμότητά του. Και τώρα περνάμε σε κάποιες από τις συνεπείς στην πολιτική ε, στην οποία αναφέρεται η μελέτη μας. Μία σύσταση που θα έκανα γενικά είναι να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε περισσότερο την έννοια της ευρωπαϊκής προσθέμενης αξίας στα εργαλεία του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Γενικά, ο αντίκτυπος του ευρωπαϊκού προπολογισμού εξαρτάται από το Πώ μπορεί να δώσει κάποια προσθέμενη αξία και έτσι έχει μεγάλη σημασία η συνέργεια με του εθνικού περιπολογισμού. Όπω βλέπουμε όμω από την υφιστάμενη βιβλιογραφία η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία δεν υπάρχει σε κάποιου από του μηχανισμού που αξιολογούνται και άρα οι συστάσει σαν χώρα αλλά και τα θεσμικά όργανα δεν αξιολογούν την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Έτσι. Καλό θα ήταν να συμφωνήσουμε σε μια στρατηγική η οποία θα ήταν πιο πολύ προσανατολισμένη στην επιχειρησιακή πτυχή. Πρέπει όμως να, σύμφωνη, να σημειώσουμε πως ε, εάν γίνει κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιβαρύνει υπέρμετρα τα κρατη Μία άλλη σύσταση που κάνουμε είναι να δούμε πιο μακροπρόθεσμα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ε, διαδικασία παρακολούθησης. Σε γενικές γραμμές η διαδικασία αυτή οργανώνεται σε αιτήσια βάση και άρα κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται η διαδικασία σε νέες συστάσεις ανά χώρα. Αυτό σε γενικές γραμμές σημαίνει πως η παρακολούθηση είναι μια απαραίτητη διαδικασία, προσανατολίζεται στα αποτελέσματα και έτσι χάνουμε κάποιες ευκαιρίες καθώς η υλοποίηση κάποιων από των συστάσεων ίσως χρειαστεί περισσότερο από ένα έτος βεβαίως. Έχει κάποια αξία η έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά δεν μπορεί να δώσει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε που χρειάζονται για την αξιολόγηση. Παραδείγματο χάρη, όταν μιλάμε για μακροοικονομικά δεδομένα για να αξιολογήσουμε την συμμόρφωση με τι ε, συστάσει, τα δεδομένα μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο αργότερα. Επίση, μια άλλη σύσταση είναι να συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε μεγαλύτερη ευελιξία του ευρωπαϊκού προπολογισμού, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων τη ε, ετήσιας ε, έρευνας για την ανάπτυξη. Γιατί μπορεί έτσι να υπάρχει περισσότερη υπευθυνότητα στον προπολογισμό, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα ίσως ε, όσον αφορά το θέμα της ευελιξίας. Οπότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα μέσα ευελιξίας, κάποιες ε, μεταφορές και την δημιουργία νέων μέσων του προϋπολογισμού που θα χρησιμοποιήσουν τα νέα κονδυλία όπως παραδείγματο χάρη το νέο, το νέο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Οπότε φαίνεται ότι σε γενικέ γραμμέ ε, και οι αρμόδιοι και οι ειδικοί ε, σύμφωνοι με αυτό. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να πούμε ότι απαιτείται πρόσοχη έτσι ώστε τα ευελικτά αυτά μέσα να μην αποδυναμώσουν την διαφάνεια και τη λογοδοσία. Και τέλο, για να τελειώσω τη σημερινή παρουσίαση, έχω και ορισμένα άλλα ζητήματα που θα έπρεπε να λάβετε υπόψη. Πρώτα απ' όλα, όπως ε, είπαμε, το τομείς προτεραιότητας ε, υπάρχουν σε τρεις κυρίως κατηγορίες. Ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μέτρα για την ανάπτυξη και άλλα. Οπότε υπάρχει γενικά η συνένεση πως υπάρχει δυνατότητα να αξιθούν οι δημόσιες δαπάνες. Κάποιες δαπάνες όμως προσπάθησαν να ποσοτικοποιήσουν τον πιθανό αντίκτυπο αυτών των ε, μέτρων και κυμαίνονται μεταξύ 3 και 10% αναλόγως του αναλόγως με το χρονικό διάστημα. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν καταλήξει σε θετική αξιολόγηση αυτών των μέτρων, επόμενη διαφάνεια, αλλά... Πρέπει να τονίσουμε εδώ πω ε, παρά το ότι αυτέ οι ανησυχίε για τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων υπάρχουν, διάφορε μελέτες έχουν θέσει διάφορα ερωτήματα για το εάν η δημοσιονομική εξυγένση και άρα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι τα καταλληλότερα. Υπάρχει επίσης το ζήτημα, όπω είπαμε, της δημοσιονομική ε, υπαναχώρηση υπαναχώρησης και το εάν μπορεί να είναι θετική για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία, ειδικά για χώρε οι οποίε αντιμετωπίζουν αρνητικέ συνθήκε. Ιδιαίτερα Κάποιοι αμφισβητούν το εάν μπορεί ποτέ η δημοσιονομική, ε, ο δημοσιονομικός περιορισμός να οδηγήσει σε ανάπτυξη. Οπότε το θέμα είναι πώς θα συνδυάσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις στην δημοσιονομική εξεγένση και τις επενδύσεις. Και φτάνουμε τώρα στο τέλος της παρουσίασής μας. Πάνω στην ώρα νομίζω. Και είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Merci, merci pour euh, cette étude et Ευχαριστούμε αυτή τη μελέτη και την παρουσίαση. Φυσικά εδώ κάνουμε ε, σκέψεις και θεωρήσεις μακροοικονομικές ε, και βεβαίως ε, αναρωτιόμαστε ποιοι είναι οι σωστοί, τα σωστά σημεία πίεσης ας πούμε για μια καλή ανταπόκριση. Ομολογώ ότι είναι περίπλοκο το ζήτημα, προκαλεί προβληματισμούς. Ε, λέτε στην εκθεσή σας ότι υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ε, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία. Κατά την άποψή σας ε, πρέπει να υπάρχει εκλογήκευση και... Ε, μια ευθυγράμμιση όσον αφορά τις κατευθύνες γραμμές ε, του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου ε, και του εξαμήνου. Ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός υποστηρίζει αρκετά τους στόχους της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης και τους αναπτυξιακούς στόχους. Δηλαδή υπάρχει αρκετός βαθμός ευελιξίας έτσι ώστε κάθε χρόνο να ε, ε, ε, κάνουμε τις απαραίτητες δράσεις. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που δεν μπορεί να διορθωθεί ή μπορείτε να φανταστείτε κάποια εργαλεία έτσι ώστε καλύτερα να ευθυγραμμιστεί η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης με την ανάπτυξη. Επίσης υπάρχουν κάποιοι νέοι δείκτες γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί όλους, νυχθημερών το σκεφτόμαστε έτσι ώστε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μπορείτε να μας δώσετε την άποψή σας ε, όσον αφορά τα μέσα που έχουμε ή μπορούμε να ε, έχουμε για να αξιολογήσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία και ποιος κατά την άποψή σας ε, έχει ε, την ε, δυνατότητα να μετρήσει αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είπατε επίσης ε, ότι μακροπρόθεσμη προοπτική θα χρειάζεται έτσι ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κατά την άποψή σας, ποια είναι ή ποια θα ήταν η ιδιώδης περίοδος αναφοράς για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματά σας καταδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο αξιολόγησης ε, της Κομισιόν ή άλλων όσον αφορά την ε, υλοποίηση των συστάσεων αναχώρα. Ε, ποια είναι η πρότασή σας έτσι ώστε να μειωθούν αυτές οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες μέλη και την Κομισιόν. Τέλος, αναφέρεστε στην ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνάς σας, πώς αξιολογείτε το ΕΦΣΑ ως νέο εργαλείο. Αυτή είναι μια πρώτη σειρά ερωτήσεων τις οποίες εγώ σας υποβάλλω και τις ε, οποίες ενδεχομένως θα μπορέσετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ καλές ε, ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Να ξεκινήσω από εκεί. Είπαμε ότι πρέπει να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες για να την αξιολογήσουμε και εδώ ειδικά θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε πιο συγκεκριμένα δεδομένα για το εάν αυτά τα έργα δημιουργούν κάποια αξία για τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι το επίπεδο της αξιολόγησης πρέπει να γίνεται από κοινού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη, αλλά με ίσως λίγο περισσότερη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε κάποιους μηχανισμούς παρακολούθησης σε γενικές γραμμές κοιτάμε το εάν ε, τα έργα ή τα κονδύλια που χρηματοδοτούν ε, εθνικά έργα ε, θα έχουν κάποια ιδιαίτερη προσθέμενη αξία σε σχέση με τα εθνικά κονδύλια. και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ακόμα αναφέρει συγκεκριμένα στη μελέτη μας. Όταν δούμε την μεγαλύτερη ευελιξία βασιστήκαμε στην υφιστάμενη βιβλιογραφία Είδαμε δηλαδή ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο Μέχρι στιγμή, δεν έχουμε δει ακόμα λοιπόν τις συζητήσεις για την μεταρρύθμιση αυτών, αλλά υπάρχει κάποια ευθυγράμμιση εδώ πέρα στα διάφορα επίπεδα προτεραιοτήτων που σχετίζονται με την αιτήσια έρευνα για την ανάπτυξη και την ανάλογη κατανομή του προπολογισμού για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν υπάρχει ακόμα μια σαφής αξιολόγηση αυτών των τομείων, αλλά η πρώτη ε, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τις δραστηριότητες της ε, ετήσιας μελέτης για την ανάπτυξη. Θα δώσω το λόγο στην, στην κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την μελέτη σας και την εξαιρετική παρουσίαση. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τα ευρήματά σας που τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα είπατε ότι με την στενή ενία υπάρχει κάποια συνέργεια μεταξύ των εθνικών και του κοινοτικού προπολογισμού αλλά με την ευρύτερη ενία είναι δύσκολο να αξιολογηθεί αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτό. Χρειαζόμαστε διαφορετική δομή του προπολογισμού που θα συνδέεται περισσότερο με τις προτεραιότητες που ορίζει η τη μελέτη για την έρευνα. Και επίσης, στις συστάσεις για την πολιτική λέτε, που τις ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, λέτε ότι χρειάζεται πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και με κάποιον τρόπο περισσότερη ευελιξία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σημαίνει αυτό ότι χρειαζόμαστε κάπως στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για αυτή την διαδικασία οικονομικής πολιτικής μήπως ε, να έχουμε πρώτα απ' όλα επταετής προοπτικές και το τι πρέπει να γίνει στα 7 χρόνια και μετά να συνδέσουμε τους επταετής στόχους με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τους Εθνικούς Προϋπολογισμούς χρειαζόμαστε και στο εθνικό επίπεδο μακροπρόθεσμες προοπτικές ε, και εθνικούς προπολογισμού για να έχουμε τη σύνδεση των στρατηγικών στόχων μέσω του προπολογισμού και από εκεί να δούμε δράσεις και έργα που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Γιατί αναρωτιέμαι πώς θα έχουμε αυτή την δυνατότητα να αξιολογήσουμε ευρύτερα τα αποτελέσματα των συνεργειών. Ευχαριστώ. Γενικά, όπως αναφέρατε, υπάρχουν συνέργειες μεταξύ του κοινοτικού προπολογισμού και των προτεραιοτήτων της ε, ε, ετήσιας έρευνας. Είναι δύσκολο εμπειρικά να αξιολογήσουμε την σχέση μεταξύ εθνικών συστάσεων και προϋπολογισμών. Δηλαδή υπάρχει κάποια αιτιώδης ε, σχέση στις αλλαγές που βλέπουμε, αλλά υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στα δεδομένα και δεν μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα των προϋπολογισμών με βάση τις ε, προτεραιότητες αυτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μετά είδαμε τις αλλαγές σε βάθος χρόνου, οποιαδήποτε αιτιώδης σχέση. Είναι δύσκολο να φανεί, ειδικά σε αιτήσια βάση, γιατί είναι τόσοι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τους προπολογισμού πέρα από τις ε, συστάσεις αναχώρα, ώστε είναι γενικά δύσκολο. Όπως είπατε, αν ε, το δούμε πιο μακροπρόθεσμα και όχι μόνο σε αιτήσια βάση, ίσως ε, διευκολυνθεί η κατάσταση, δηλαδή να έχουμε περισσότερα δεδομένα για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τις αλλαγές σε βάθος χρόνου. Τώρα, επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα το οποίο δεν απάντησα. Μιλάμε για τον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Είναι δύσκολο να δούμε αν θα είναι τρία-τέσσερα χρόνια, αλλά προτείνεται έναν ορίζοντα επταετίας. Αυτό ίσως μπορεί να βοηθήσει να αξιολογήσουμε γενικά αν είναι ευθυγραμμισμένες οι προτεραιότητες. Μήπως όμως εδώ προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. γιατί ποια μπορεί να είναι η επίπτωση ενός προπολογισμού που αντιπροσωπεύει το 1% του ΑΕΠ, Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, δηλαδή ένα πεντηκοστό του μέσου όρου των εθνικών προϋπολογισμών, πλαισιωμένο σε ένα πλαίσιο 7 ε, ετών, με κατανομή στα κράτη-μέλη ε, της τάξης του 70%, ε, σαν στρατιωτικά ταμεία, σαν ταμεία συνοχή, σαν γεωργικά ταμεία κτλ. Πώς. Ε, ε, είναι άκαμπτο εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να λάβει υπόψη την, πραγματικά την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης. Έχετε επίσημη άποψη γι' αυτό, δόκτωρ. I Δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. Εμείς βλέπουμε τις προτεραιότητες, αν είναι ευθυγραμμισμένες ε, και αν ε, οι συστάσεις αναχώρα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις ε, αρχές. Δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα μακροχρόνια προοπτική σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς. Ναι, αλλά δεν χρειάζεται προϋπολογισμός της Ευρωζώνης. προπολογισμό λοιπόν τη Ευρωζώνη, ακριβώς έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αναέτος και λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ε, προϋποθέσεις ε, και τις περιπτώσει που ισχύουν σε κάθε χώρα. Ελήψη αυτού θα έχουμε απλώς έναν άκαμπτο μηχανισμό που στην ουσία θα εξακολουθήσουν να, έχουν, να είναι ασύ, μια, μια ασημαντότητα από πλευράς προπολογισμού, δηλαδή 1%. Δηλαδή 7 χρόνια πριν να ξέρουμε τι, ε, ε, τι θα πρέπει να πάρει κάθε χώρα ή τι αρμόζει σε κάθε χώρα, αυτό είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου. Ne, ε, κοιτάξτε, ε, ε, σπάστε λίγο τα δεσμά της ε, συμβατότητας. Μην μιλάτε με αυτήν την πάγια διατύπωση. Είπα ότι όντως υπάρχει, όντως είναι και μου άποψη, ότι υπάρχει μία ακαμψία λόγω αυτής της εφταετούς περίοδου. Αλλά, πώς να σας το πω. Εάν πρέπει κανείς να ανταποκριθεί σε νέες ε, προϋποθέσεις και απαιτήσει. Έστω και αν είναι μικρός ο προϋπολογισμός σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ε, έστω και αν υπάρχει λέω αυτή η ακαμψία, θα μπορούσαν να κινητροδοτηθούν κάποιες επενδύσεις. Δηλαδή λέω ότι μπορεί η όλη διαδικασία να είναι ε, άκαμπτη σε αυτή τη μεγάλη χρονική περίοδο, αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο όσο το να τετραγωνίσει κανείς τον κύκλο. Ίσως η Κομισιόν να μας πει κάτι. Ίσως η Κομισιόν λοιπόν να πάρει το λόγο πρώτα απ' όλα να μας πει ποια είναι η άποψη της Κομισιόν όσον αφορά αυτά τα στοιχεία. Ποια είναι η εκτίμηση της ε, Κομισιόν όσον αφορά την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και τις ε, προσαρμογές ε, που έχουν γίνει Δηλαδή θεωρεί ότι υπάρχει έτσι επιχειρησιακή κίνηση ή ε, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι καταφέρνουν. Τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται από τις χώρες μήπως ε, θα πρέπει να ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα έτσι ώστε να αυξηθεί η συγκρισιμότητα. Καλό θα ήταν να έχουμε ε, μία στάνταρ παρουσίαση των προϋπολογισμών έτσι ώστε να έχουμε κοινή γλώσσα γιατί τώρα ο καθένα λέει τα δικά του και οι διαφορέ είναι μεγάλε. Πώ μπορεί να είμαστε στην ίδια κοινότητα εάν δεν μιλάμε με, την ίδιο, με τις ίδιες λέξεις, με το, την ίδια ορολογία, με το, με το ίδιο συντακτικό. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η οργανική ανάγκη η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και την Επιτροπή των Προπολογισμών για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να διοργανώσει, να ζητήσει την ε, διεξαγωγή αυτής και να ευχαριστήσω και τον Δ. Χαφνέρ για την παρουσίαση που έκανε. Ε, θα ξεκινήσω την ε, απάντηση από την της Επιτροπής κάνοντας κάποιες αρχικές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό της Ένωσης και το πώ αυτό περιγράφεται στη μελέτη. Και από εκεί και μετά θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ, η οποία σίγουρα θα έχει κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά την ε, ετήσια επισκόπηση τη ανάπτυξη και το πώ αυτή σχετίζεται με του ε, εθνικού προπολογισμού. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω τέσσερα σύντομα σχόλια σε ό,τι αφορά τον ετήσιο προπολογισμό. Τον προπολογισμό της Ένωσης, όπως περιγράφεται στην παρούσα μελέτη. Ε, εκτιμούμε καταρχήν το γεγονό ότι η μελέτη αναγνωρίζει το ότι ένα μεγάλο τμήμα του προπολογισμού της Ένωσης προσανατολίζεται προς τις επενδύσεις, ακριβώς για τη δημιουργία της, ε, των θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης. Η κατά συνέπεια ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της αιτήσιας επισκόπηση ανάπτυξης. Και πράγματι αναγνωρίζει η μελέτη ότι μέσω των γραμμών ένα α και ένα β του προπολογισμού γίνονται ακριβώς αυτές οι ε, επενδύσεις και οι εν λόγω γραμμές έχουν αυξηθεί σε ό,τι αφορά τα κονδύλια τους, δηλαδή μέσα στα τελευταία χρόνια. Επίσης αναφέρεται σωστά η μελέτη στον αυξανόμενο ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και εδώ ενδεχομένω καλό θα ήταν να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονό ότι η μελέτη αναφέρεται στο ότι ε, το ΕΦΣΙ ανταποκρίνεται στο 10% των ε, ε, πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ε, στο πλαίσιο της, του συγκεκριμένου κεφαλαίου του προπολογισμού. Αλλά βέβαια αυτό αποτελεί μόνο ένα ε, τμηματικό αν θέλετε ε, αντίκτυπο της αξιοποίηση του ΕΦΣΙ γιατί έχει γενικά μοχλεύσει κεφάλαιες τάξεις των 200 δις ήδη το ΕΦΣΙ. Τώρα σε ό,τι αφορά τις συνέργειες μεταξύ προπολογισμού της Ένωσης και εθνικών προϋπολογισμών. Πράγματι αναφέρεται εδώ ότι ε, αυτός ο συντονισμός αν θέλετε γίνεται μέσω των κοινών απαιτήσεων σε χρηματοδότηση και μέσω των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Ωστόσο οι συνέργειες κατά τη δική μας άποψη δεν σταματούν εδώ και να σας δώσω και ένα παράδειγμα εδώ ε, προφανές το οποίο γνωρίζουμε καλά όλοι και αυτό είναι ε, η ανταπόκριση του προπολογισμού στην ε, κρίση του ε, προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Δηλαδή, μέσω εδώ των συνεργειών των εθνικών προπολογισμών και του προπολογισμού της Ένωσης, καταφέραμε να ανταποκριθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της σε αυτήν ε, την τεράστια νέα πρόκληση που βρήκαμε μπροστά μας και την οποία δεν θα ήταν σε θέση τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αν ήταν ε, μόνο του δηλαδή την υποστήριξη της Ένωση. Από εκεί και μετά ένα τρίτο σχόλιο ε, που θα ήθελα να κάνω αφορά την προστιθέμενη αξία του προπολογισμού της Ένωσης. Όπως αναφέρεται ε, και στη μελέτη, πράγματι είναι πολύ μικρός ο προπολογισμός της Ένωσης και ανταποκρίνεται μόνο στο 2% των εθνικών προπολογισμών κατά μέσο ώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς ως επροβολούς της Ένωσης να οριζόμαστε ως προς την αξία του δηλαδή με βάση την προστιθέμενη αξία που έχει για την Ένωση. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό επενδύοντας σε έργα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί σε διαφορετική περίπτωση. για παράδειγμα ένα από τα έργα, αν θέλετε, τα κυριότερα έργα, όπως για παράδειγμα το στην Ευρώπη, το η διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη ή το Erasmus δεν θα ήταν δυνατό να έχουν υλοποιηθεί χωρί τα κονδύλια του προβληματισμού τη Ένωση. Άρα λοιπόν σε τέτοιου είδου έργα να αναφερόμαστε, τα οποία δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί, δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί τόσο γρήγορα αν δεν υπήρχαν τα κονδύλια της Ένωσης. Και από εκεί και μετά υπάρχουν, πέραν δηλαδή αυτών των έργων, Είμαστε πεπισμένοι ότι μέσω του προπολογισμού της Ένωσης ε, χρηματοδοτούμε έργα υψηλότερης ποιότητας από αυτά που θα είχαν χρηματοδοτηθεί από τους εθνικούς προπολογισμούς. Και εδώ αναφέρομαι ειδικότερα στο Horizon 2020, καθώς μέσω εδώ της, της, ε, συγκέντρωσης, αν θέλετε, ε, των πόρων, μέσω κοινών προκήρυξων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε όλα τα κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ήμασταν θέση να αυξήσουμε τόσο την ποιότητα των προσφορών αλλά και να συγκεντρώσουμε και υψηλότερη χρηματοδότηση από ότι αυτό θα ήταν δυνατό στο πλαίσιο των ε, εθνικών προϋπολογισμών. Ένα τελευταίο σχόλιο που δώσω το λόγο στη συνάδελφου από το ΕΚΘΗΝ είναι η ε, ευελιξία. Δηλαδή, μέσω της ευελιξίας του προπολογισμού της Ένωσης, ήμασταν σε θέση να ανταποκριθούμε σε μία σειρά από νέα προβλήματα και νέες προκλήσεις. Η μελέτη αναφέρει εδώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αλλά και την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και πράγματι και αυτές οι δύο νέες πρωτοβουλίες ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθούν μέσω της ευελιξίας που προβλέπεται στον προπολογισμό της Ένωσης. Άρα λοιπόν το πόρισμα της μελέτης ε, που αναφέρει το ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και να υπάρξει και η ε, από την πλευρά του Συμβουλίου με την συνένεση του Κοινοβουλίου τη ε, ε, ενδιάμεσης αναθεώρηση, είναι σωστό. Γιατί η ενδιάμεση αναθεώρηση δεν θα είχε λάβει χώρα χωρί την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και είναι αυτή η οποία παρέχει την προστιθέμενη ευελιξία στον προπολογισμό στα πλαίσια ακριβώς των υπολοιπόμενων 3,5 ετών του παρόντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που ενδεχομένως θα ανακύψουν ε, ε, μέχρι ακριβώς την ολοκλήρωση αυτού του πολυνοητού σε δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά από την πλευρά μου πρόεδρε και θα δώσω τώρα το λόγο και στη συνάδελφο από τη Γενική Διεθνήση ΕΚΦΙΝΑ. Ναι, λέω σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε, για την παρουσίαση αυτή και για τα πολύ προσφυγή ερωτήματα που θέσατε. Ε, συμφωνώ και εγώ μαζί σας ως προς το ότι δηλαδή θα πρέπει λίγο να θέσουμε το γενικότερο πλαίσιο της όλης συζήτησης, δηλαδή ε, ποιο είναι το, το φάσμα θέλετε, που καλύπτει ο ε, προπολογισμό ε, με βάση και τη σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε χθε γιατί αυτό θα μας βοηθήσει αφού πρόκειται για το ζήτημα της προσθέμενης αξίας του προβλογισμού της Ένωσης όταν κάνουμε τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του πολυδιεπτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δηλαδή οι γενικές γραμμές πολιτικής είναι εκείνες οι οποίες ε, κατευθύνουν αν θέλετε τον προπολογισμό προς την κατεύθυνση της ε, υποστήριξης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς οι οποίοι για παράδειγμα να έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να μην σχετίζονται άμεσα με την αναπτύξη και την ε, δημιουργία θέσεων εργασία. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώ εδώ πού στοχεύει ο προπολογισμό. Επίση, η τελική έκθεση τη ομάδα υψηλού επίπεδου για του ίδιου ε, πόρου ήταν πολύ σημαντική γιατί υπήρξε εκεί μια σύσταση για ακριβώ την ε, ε, την αύξηση της ε, συνέργειας μεταξύ των εθνικών προπολογισμών και ε, της, του εθνικού του προπολογισμού της Ένωσης και η ενόχως σύσταση μπορεί να χωριστεί σε τρία τμήματα. Δηλαδή, καταρχήν για να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες θα πρέπει να εντοπίσουμε τους τομείς εκείνους όπου έχει νόημα ακριβώς να αναλυφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό. Και ένα σχετικό, για σας ξαναλέω ότι το έγγραφο με κάποιες σκέψεις ε, δημοσιεύτηκε χθε, ο οποίο δηλαδή εδώ αναφέρει κάποια σενάρια και κάποιες ε, ιδέε. Κάτι το οποίο βέβαια να μην αφορά ενδεχομένω άμεσα την Επιτροπή Πολυλογισμών, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και μετά, προκειμένου να υπάρχει αυτή η ε, κάθετη συνοχή, αυτό το vertical coherence, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, συμμόρφωση μεταξύ πολιτική και των προπολογισμών. Δηλαδή, αν δούμε για παράδειγμα την πολιτική σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, θα δούμε ότι αν έχουμε μια τέτοια φιλόδοξη πολιτική, ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε και του επαρκεί πόρου ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, επειδή δεν υπάρχουν πάντοτε αυτά τα κονδύλια, ε, γι' αυτό χρειάζεται και ευελιξία στον προπολογισμό. Και ακριβώς αναφέρομαι στο μεταναστευτικό γιατί ε, δεν εξετάζεται ω τέτοιο στο πλαίσιο τη ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη. Μπορεί δηλαδή μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε περισσότερη ανάπτυξη, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη ω τέτοιο. Και ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα και αυτό με το ζήτημα της κάθετης ε, συνοχής, είναι η σχέση μεταξύ προπολογισμού της Ένωσης και εθνικών προπολογισμών με βάση τις εθνικές πολιτικές. Γιατί εάν δούμε ποιο είναι ε, το μέγεθος του προπολογισμού της Ένωσης, είναι μόνο το 1% του ΑΕΠ ε, της Ένωσης και 2% του μέσου των εθνικών προπολογισμών. Άρα λοιπόν η προστιθέμενη αυτή αξία του προπολογισμού της Ένωσης καθορίζεται από τα κράτη-μέλη. Εκείνα δηλαδή ε, είναι ε, αυτά που θα πρέπει να αποφασίσουν πού χρειάζονται υποστήριξη ως ένα πρώτο βήμα, αλλά και από εκεί και μετά θα πρέπει ο προπολογισμό της Ένωση να χρησιμοποιείται για να προωθούνται μεταρρυθμίσει στου ε, τομεί εκείνου των κρατών μελών όπου χρειάζεται να υπάρξει, να αναλυφθεί δράση. Και εδώ αναφερόμαστε βέβαια και σε επενδύσει ή εν περιπτώσει άλλα είδη δαπάνης. Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο συνέργειες μεταξύ ε, εθνικών προπολογισμών και ε, κονδυλίων Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να, να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στον τομέα της ε, έρευνας και της ανάπτυξης, εδώ να πούμε ότι η Ένωση δαπανά ε, μεγάλο όγκο κονδυλίων, αλλά οι ε, εθνικοί προπολογισμοί προβλέπουν ακόμα περισσότερα κονδύλια. Οπότε λοιπόν ακριβώ στο πλαίσιο τη ενδιάμεση αναθεώρηση και στο πλαίσιο του καθορισμού των γενικών προτεραιοτήτων θα μπορούσε ακριβώ να εξεταστεί το ενδεχόμενο του να αυξηθούν τα σχετικά κονδύλια για να υπάρξουν περισσότερε ακόμα συνέργειε. Προφανώ δεν θα είναι ποτέ δυνατό να χρηματοδοτηθούν πλήρω σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολιτικέ έρευνα και ανάπτυξη, αλλά σίγουρα μπορεί να υπάρξει κάποια υποστήριξη. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πλαίσιο έτσι, της, ε, της συνοχής ε, μεταξύ ε, προπολογισμού τη Ένωση και εθνικού προπολογισμού. Και σε ό,τι αφορά τώρα κάποια επιμέρους στοιχεία της παρουσίασης που ακούσαμε. Από ό,τι κατάλαβα, οι συστάσεις αναχώρα εξετάστηκαν για τα τελευταία ε, χρόνια και θεωρήθηκε ότι ήταν σχετικά σταθερές αν θέλετε οι συστάσεις. Αλλά οι συστάσεις αναχώρα εκπονούνται από το 2011 και ε, με τη νέα Επιτροπή ε, ξεκίνησε και μια ανακατεύθυνση αν θέλετε, μια νέα στόχευση των συστάσεων αναχώρα η οποία ενδεχομένως δεν έχει ληφθεί πλήρως υπόψη στην μελέτη. Και βέβαια υπήρξαν και αντίστοιχε αλλαγέ στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη, η οποία απηχεί δηλαδή τι αλλαγέ τη τάση αναχώρα. Και εδώ αναφέρομαι ειδικότερα στι επενδύσει. Ακριβώ γιατί η ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη και η ιδιαίτερη έμφαση που έδωσε στις επενδύσει, οδήγησε και στις αντίστοιχες συστάσεις αναχώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ε, εκτέλεση των, ε, ή την, την υλοποίηση των συστάσεων αναχώρα, ε, να σας πω ότι έχω δει διάφορες συστάσεις και πραγματικά τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ διαφορετικά. Ε, δηλαδή δεν θα μπορούσε ποτέ να, να πει κανείς ότι είναι πάντοτε ίδια τα αποτελέσματα των συστάσεων. Γιατί εδώ δεν έχουμε ε, μαύρο ή άσπρο. Δηλαδή τι λέμε όταν εννοούμε ε, ότι δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως μια σύσταση χώρα. Η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για, το, για, το, για την μη εφαρμογή. Το κοινοβούλιο της χώρας ε, ήταν ε, υπεύθυνο. Οπότε, ε, εντάξει, ακριβώς για αυτούς τους λόγους δεν υπάρχει διαξιολόγηση της εφαρμογής της σύστασης από την Επιτροπή και από το εκάστοτε κράτος μέλος. Ε, και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τον ετερογενή χαρακτήρα των ε, ε, των προτεραιοτήτων, δηλαδή του πώ ε, καθορίζονται οι προτεραιότητε σε ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη και το πώ αυτέ τελικά μεταφράζονται τόσο εισαγωγικών ε, στα σχέδια των κρατών και στο επίπεδο των συστάσεων αναχώρων Να σα πω εδώ ότι και πάλι υπάρχει ένα αντιστάθμισμα. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν κάποιε γενικέ προτεραιότητε που καθορίζονται στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη, αλλά από εκεί και μετά οι ιδιαίτερε ανάγκε του κάθε κράτου μέλου διαφοροποιούνται φυσικά μεταξύ του. Οπότε, ίσω είναι θετικό το γεγονός ότι ακριβώς δεν μεταφράζονται αυτές οι γενικές αρχές ε, απευθεία σε συστάσει αναχώρα. Γιατί υπάρχει ακριβώ και εδώ μια ανάγκη περαιτέρω ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι προτεραιότητε τη επισκόπηση ανάπτυξη έχουν νόημα ή είναι, είναι χρήσιμες για το εκάστοτε κράτος μέλος. Ε, δηλαδή, ναι, λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή τη διαφορά, αν θέλετε, την απόκριση, αλλά από την άλλη πλευρά ενδεχομένω αυτή η απόκληση να είναι θετική για να ληφθούν υπόψη οι του κάθε Αυτά λοιπόν ε, ω κάποια σχόλια σε σχέση με αυτή την παρουσίαση και ελπίζω να απάντησα σε κάποια από τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω ακόμα όσον αφορά την ε, ομογενοποίηση, ε, την τυποποίηση και την παρουσίαση των δημοσίων προπολογισμών των κρατών μελών. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε προοδεύσει πολύ, έχουμε κάνει πρόοδους στο παρελθόν όσον αφορά την τυποποίηση των δημοσιονομικών δεδομένων και νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πλέον ε, τυποποίηση και ομοιογενή παρουσίαση στα κράτη-μέλη. Ευελπιστούμε ότι και αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε τώρα είναι να επιτύχουμε το ίδιο, τον ίδιο βαθμό ομοιογενοποίησης ε, και τυποποίησης ε, και σε άλλες μορφές δαπανών. Εάν καταφέρνουμε ας πούμε τους ε, δημόσιους λογαριασμούς να τους παρουσιάζαμε με τον ίδιο τρόπο θα ήταν ήδη πάρα πολύ καλό. Η, εν πάση περιπτώσει πάντως είναι ο, ε, ένας τομέας στον οποίο ε, πρέπει να κινηθούμε και να προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος. Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Η κυρία Μάιτιτς. Ευχαριστώ. Πραγματικά θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπατε και ε, κατανοώ την απάντηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, τυποποιημένες σειρές δεδομένων έτσι ώστε η επιτήρηση να είναι καλύτερη. Ας πούμε το National Mountain Fund έχει ε, δικές τους, ε, έχει συγκεκριμένο μορφότυπο για τα στοιχεία και για τα δημοσιονομικά και για τα άλλα, αλλά έχουν και λειτουργικές ε, ε, ταξινομήσεις ε, και μετά συνεδριά, συγγνώμη, συγκρίνουν τις χώρες ανάλογα με αυτά τα λειτουργικά δεδομένα. και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προγράμματα και ποιοι είναι οι στόχοι επί των οποίων θέλουμε να έχουμε ε, συγκρίσιμα στοιχεία και ε, ε, να προσαρμόσουμε λοιπόν τον ευρωπαϊκό προβληματισμό και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και επίσης, λέει ο Πρόεδρος, πρέπει να πούμε ότι αυτή η διαφοροποίηση, το κενό ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές είναι τέτοιες που ξεκινάμε ας πούμε ένα πολυετές πλαίσιο επταετές και, και στις πρώτες, τα πρώτα δύο χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Ε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι τόσο και προγράμματα τόσο περίπλοκα που δεν μπορεί να οικειοποιηθεί των κονδυλίων και των πόρων ο υπεύθυνο ε, και επομένως ε, αργεί πάρα πολύ να κινητοποιηθεί το πρόγραμμα. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε λοιπόν. Θα δώσω τον λόγο στον δόκτωρα Μάρκο Χάφνερ, ε, ο οποίος ε, ε, θα κάνει με κάποιες τελικές παρατηρήσεις και ελπίζω να μου εμφυσίσει κάποιο ενθουσιασμό εμένα που είμαι ο εισηγητής, γιατί μέχρι τώρα δεν το είδα. Λοιπόν, έκανα τις ερωτήσεις μου. Ενθουσιάστε με τώρα κύριε. So your question is what the value added of this study is. Το είναι ποια είναι η προσθέμενη αξία αυτής της μελέτης. Όχι, τη έκθεση που μου ζητούν ε, να κάνω κάθε χρόνο. Ε, ε, θέλω να ξέρω εάν χρησιμεύει σε κάτι και σε τι. To do it every year. C'était un rapport ε, κάνω μια έκθεση για, για το ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο και νομίζω ότι είναι περισσότερο σε δουλειά να βρισκόμαστε παρά ε, να δίνει προστιθέμενη αξία. Of, αξία. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι ε, έχει νόημα να γίνει τη διαδικασία κάθε χρόνο, αλλά δεν έχουμε αξιολογήσει την αξία της έκθεσης αυτής στη μελέτη μας. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Θα τη μελετήσω θα την ξεψαχνίσω, θα την ξεκοκαλίσω, σας το υπόσχομαι αυτό και θα δω εάν πραγματικά υπάρχει κάποια σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αν είχαμε ε, προπολογισμό της Ευρωζώνης θα ήταν πολύ χρήσιμο. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους και περνάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο μάλιστα αναφέρθηκε και εν παρόδο ε, στην προηγούμενη συζήτηση. Μεταρρύθμιση συστήματος ιδίων πόρων. Έχουμε δύο εξαίρετους εισηγητές, τον κύριο Λεβαντόφσκι και τον κύριο Ντεπρέ που ξεψάχνησαν την έκθεση της ομάδας Μόντι και που ε, θα μας ε, ε, που θα πάρουν τον λόγο. Ο κύριος Ντεπρέ θα ξεκινήσει. Όχι, ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ. Το έγγραφο εργασίας ήταν το εύκολο της εργασίας που έκανα με τον Ζεράρ Ντεπρέ στην προσπάθειά μας να βρούμε θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σύστημα των ίδιων πόρων. Ε, το έγγραφο αφορά την ιστορία και την εξέλιξη του συστήματος των ιδίων πόρων. Υπογραμμίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον υπογραμμίζει δεόντως, γιατί το Κοινοβούλιο ε, πάντοτε ε, ενθαρρύνει ε, την μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχουν συμπεριληφθεί επίσης και κάποια στοιχεία σκέψης, ένα ε, ερωτηματολόγιο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες αρχές οι οποίες έχουν εκφραστεί. Ε, κάποια στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών όσον αφορά ε, τα δημοσιονομικά και τη σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία. Μετά έχουμε ένα επόμενο στάδιο το οποίο είναι μεικτό και είναι πιο, λίγο πιο δύσκολο, αφορά το χρονοδιάγραμμα της έκθεσής μας, γιατί εμείς ε, Μπαίνουμε σε αμφιλεγόμενη ε, έτσι, διάσταση όταν μιλάμε για τη θέση του Κοινοβουλίου ε, και όταν προσπαθούμε να περάσουμε τη θέση αυτή στην παρούσα κατάσταση. Ε, το το όραμά μας είναι αυτό του Ελέν Λαμασούρ, δηλαδή ότι κάθε ε, ευρώ το οποίο χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, δημιουργεί αποταμίευση, να δημιουργεί επενδύσεις, ε, αλλά αυτό ακόμα δεν το έχουμε επιβεβαιώσει. η συζήτηση για, του, για τους ίδιους πόρους και τις μεταρρύθμισης των υφισταμένων οικονομικών συστημάτων στην ουσία ε, είναι, υπόκεινται μάλλον στην πολιτική βούληση και η ετοιμότητα ε, τροποποίησης ε, των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στο reflection paper της Κομισιόν το Brexit φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά το τμήμα των δαπανών, αλλά ε, ενδεχομένως ε, μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την μεταρρύθμιση ε, του συστήματος των ιδίων πόρων, γιατί μέχρι τώρα πάντα λέγαμε, αναφερόμαστε στις επιστροφές προς το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι στην μεταρρύθμιση. Είναι σαφές ότι ο Ζεράρ και εγώ θα πρέπει ε, να δουλέψουμε μαζί με την ε, συνάδελφο Τομά και τον συνάδελφο Όλμπρεχτ. Αυτό που δεν είναι σαφές και μάλιστα είναι και αμφιλεγόμενο είναι αυτό που συζητήθηκε και στους συντονιστές, δηλαδή εάν και κατά να, θα πρέπει να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να το προσαρμόσουμε στην παρουσίαση ε, της Κομισιόν έτσι ώστε να ε, ταυτιστούν χρονικά ε, οι προτάσεις ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οπωσδήποτε να ενθαρρύνουμε σαφώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναπροσπαθήσει να μεταρρυθμίσει το σύστημα ιδίων πόρων. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Γιάννους. Ο Ζεράρ Ντεπρέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα μία αποσαφήνιση σε σχέση με την Ιζαμπέλ αλλά δεν είναι εδώ, ε, γιατί είπε το πρωί ότι οι δύο συνεισηγητές για το πολιετές ε, πλαίσιο ε, ήταν ε, ήταν λίγο πιο πίσω χρονικά. Ε, ε, αυτό νομίζω ότι δεν είναι αρκετά σωστό, γιατί το δικό μας έγγραφο αναφέρεται σε καθαρά πραγματικά περιστατικά και ορίζουμε το πλαίσιο εντός των οποίων θα κινηθούν οι διαδικασίες. Υπενθυμίζουμε λοιπόν το νομικό πλαίσιο, δηλαδή πώς ε, αιτιολογούν τα άρθρα των συνθήκων την, το αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζουμε ε, κάποιες συγκεκριμένες ιδέες έτσι ώστε να τις κατανοήσουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ασθενή μνήμη. Επίσης αφιερώνουμε ένα τμήμα στην εξέλιξη του συστήματος των ιδίων πόρων καθώς επίσης και την, ε, το ποσό που τους αναλογεί, το τμήμα που τους αναλογεί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τα προβλήματα του υφισταμένου συστήματος που ε, αιτιολογεί εν μέρη και την ανάγκη μεταρρύθμισης. Ο κύριος Λεβαντόφκη ε, ήταν πολύ διακριτικός όσον αφορά την παράγραφο αυτή. Εμείς υπενθυμίζουμε εν περιπτώσει και τις πρόσφατες ή σχετικά πρόσφατες προτάσεις οι οποίες έγιναν είτε μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου είτε μετά από πρωτοβουλία της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων. Υπενθυμίσουμε επίσης την πρόταση του Ελένα Μασούρ το 2007. Υπενθυμίζουμε και το λέω εγώ γιατί ο ενδιαφερόμενος θα δυσκολευόταν να το κάνει. Αναφερόμαστε εις ε, το περιεχόμενο του νομοθετικού ε, ε, πακέτου που παρουσίασε ο Σλάνθος Λεβαντόφσκι το 2011 και επίσης κάνουμε μια σημαντική ανάλυση της ομάδας Μόντι. Η ομάδα Μόντι, κατά την άποψή μου, είναι στρατηγικής ε, σημασίας ε, για την ε, διαδικασία που κάνουμε και τη διαδικασία που ακολουθούν και όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Πρώτον, γιατί ήταν διοργανικό και τα συμπεράσματα και το περιεχόμενο είχαν συζητηθεί από τους εκπροσώπους των τριών θεσμικών οργάνων και είναι τρία τα σημαντικά συμπεράσματα ανεξάρτητα ε, από το γεγονός ότι ε, ζητούσαν τροποποίηση του συστήματος ιδίων πόρων. Πρώτον, καθορίζει ε, κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να εκτιμήσουμε τη σημασία των ιδίων πόρων με μια σειρά άλλων κριτηρίων που δείχνει ποιες είναι οι κατηγορίες οι οποίες είναι πιο καλές και ποιες πλέον ενδεικνυόμενες. Επίσης λέει ότι ένας μηχανισμός ιδίων πόρων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ε, υποστηρικτική της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και εκεί αναφέρει δύο στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά την ολοκλήρωση τελειοποίηση της ενιαίας αγοράς σε βάση της οποίας σχετίζει κάποια στοιχεία των ιδίων πόρων δυνητικών νέων με νέους δυνητικούς ιδίους πόρους και με το σύστημα της ενεργειακής μετάβασης στα πλαίσια της καταπολέμησης της κλιματικής ε, αλλαγής. Εν πάση περιπτώσει, τα ερωτήματα τα οποία εμείς ε, θέτουμε ε, αφορούν την, τις λύσεις και πώς αυτές μπορούν να γίνουν πιο επιχειρησιακά υλοποιήσιμες. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά λιγότερο το Εθνικό Κοινοβούλιο και περισσότερο τα εθνικά ε, κράτη, τα οποία είναι πολύ πιο μοιρασμένα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων. Η ερώτηση είναι, θέλετε ένα νέο σύστημα το οποίο, ιδίων πόρων το οποίο θα αυξήσει ε, την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θέλετε να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο. Ε, δεύτερη ερώτηση το ζήσμα των ιδίων πόρων θα πρέπει ε, να ε, ε, αυξηθούν ή θα πρέπει να μειωθούν. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τη σωστή μεταρρύθμιση θα πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα Έχουμε και μία τρίτη κατηγορία ερωτήσεων σχετικά με τις ενδεχόμενες διορθώσεις, έστω και αν διατηρήσουμε το σύστημα του GMI υπάρχει ένα φαινόμενο ιδιαίτερο, δηλαδή η ε, ε, κατακεφαλή συμβολή ε, και το κατακεφαλή ΑΕΠ Ε, που συμβάλλουν στον προϋπολογισμό δεν έχουν απαραίτητα ε, ψηλότερο κατακεφαλή εισόδημα από τις χώρες οι οποίες δέχονται ε, τις, την υποστήριξη από τον προϋπολογισμό. Επομένως το ζήτημα του καθορισμού ε, του ΑΕΠ, ε, βάσει του οποίου καθορίζεται και η συμβολή ε, βάσει του ΑΕΠ, θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθεί. Συμφωνείτε επίσης ότι οι κατηγορίες των ή η κατηγορία των ιδίων πόρων θα πρέπει να ενταχθούν στην, στην στρατηγική της μεγάλης αγοράς στην οποία είχε καταλήξει η έκθεση Μόντι. Ε, και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ενδεχομένως μια νέα, ένα νέο πόρο ΦΠΑ και κυρίως ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί ε, μια νέα φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Συμφωνείτε λοιπόν να επαναστοχοποιηθούν, να επανεστιαστούν μάλλον αυτοί οι ίδιοι πόροι. Και επίσης εάν αποφασίσουμε ε, να έχουμε ένα είδος ε, τροποποιημένων ιδιοπόρων ή πολλούς τροποποιημένους ίδιους πόρους ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει επαναστόχευση και επανεστίαση γιατί όλες οι χώρες δεν βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια κατάσταση σε σχέση με το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο είδος ιδίου πόρου και επομένως για λόγους δικαιοσύνης και ισοδίκαιας αντιμετώπισης θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Ε, εν πάση περιπτώσει να σας πω ότι εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε ε, με ευφύ τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις ενδείξεις σας και τις προτάσεις σας και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε εν πάση περιπτώσει την ε, ε, διαρκή σας υποστήριξη. Ευχαριστούμε. Ζεγάρ, λέει ο Πρόεδρος, μας δώσατε κάποιες ιδέες σχετικά με τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων, ήδη ε, οι πόροι που ε, έχουν στόχο ε, την μείωση της εξάρτησης των κρατών μελών και όχι βέβαια τη δημιουργία επιπλέον οικονομικού άκθους. Ευχαριστώ κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Λεβαντόφσκι και Ντεπρέ για αυτό το... Ε, για αυτό το έγγραφο εργασία. Εγώ είμαι εισηγητή στην Κομάγκρη για το θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό βεβαίω για το πρόγραμμα ε, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ε, κυρίω μετά από το Brexit. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαρκώ ζητά ε, ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτείται πλήρω και εξ ολοκλήρου από το σύστημα ιδίων πόρων όπω εξάλλου αναφέρεται και προβλέπεται στι συνθήκε. Και επίση έχει καθορίσει και τα όρια και το, των, του υφισταμένου συστήματος ιδιών πόρων που είναι ε, ιδιαίτερα περίπλοκο, ακατανόητο για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες που εν τέλει είναι αυτοί που βάζουν τα λεφτά τους ε, και καθόλου συγκρίσιμο. Η παρούσα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 74% στον παρόντο προπολογισμό λέω προέρχεται από εθνικές συμβάσεις 11% από τον ΦΠΑ και έχει οδηγήσει σε, στη δημιουργία πολλών ασαφών και σίγουρα ε, αδιαφάνων μηχανισμών ε, αντιστάθμισης. Πράγμα που κάνει ιδιαίτερα περίπλοκη τη διαδικασία του ετήσιου προπολογισμού. Χρειαζόμαστε νέου ίδιου πόρου ε, σε ένα ε, πλαίσιο πιο ε, σαφέ και που θα είναι σαφέστερα συνδεδεμένοι οι πόροι αυτοί με πολιτικέ ευρωπαϊκέ οι οποίε θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει επίση να ξαναδούμε λίγο το συσχετισμό εθνικού ΑΕΠ και ευρωπαϊκού προπολογισμού και να προβλέψουμε του διορθωτικού ευρωπαϊκούς ε, μηχανισμούς ε, με την ευκαιρία και κιόλας ε, του Brexit. Επίσης, το θέμα των ιδίων πόρων έχει ήδη συζητηθεί από την ομάδα υψηλού επίπεδου του οποίου προείστατο και στο οποίο προείδρευε ο, κύριος Μόντι είχε αναφερθεί επίσης και σε άλλα στοιχεία μεταρρύθμιση του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφορές ηλεκτρική ενέργεια, ψηφιακή ε, τεχνολογία, ε, το ΕΒΙΣ, το αντίστοιχο του, του Αμερικανικού ΕΣΤΑ, εν πάση περιπτώσει, είχε αναφέρει πολλά συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την χρηματοδότηση των νέων προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μετανάστευση, προσφυγικό, μη τρομοκρατία κλπ. Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται και στο reflection paper του Επιτρέπου Έτιγκερ που ε, ε, ε, πραγματικά είναι έτοιμοι να πάρουν χρήματα, να κάνουν εισβολή στη γεωργική πολιτική και στην πολιτική συνοχή σε πράγμα το οποίο εμείς δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να ξεκινήσει από το Κοινοβούλιο αυτή η ιδέα η οποία θα πρέπει να προωθηθεί και προς, όλες τις προς όλα τα άλλα όργανα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Πολύ σύντομα. Το θέμα των ιδίων πόρων είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως ε, θα αποτελέσει και μία από τις ε, κυρίαρχες ε, μάχες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την εργασία τους γιατί είναι πολύ αποσαφινιστική μας μας δείχνει από πού ξεκινάμε, πού θέλουμε να πάμε ή εν πάση περιπτώσει ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε έτσι ώστε να βρούμε το δρόμο μας προς το μέλλον. Ε, είναι ευρία η, ευρύ το έργο τους, είναι ευρία η αναφορά στους ε, ίδιους πόρους. Νομίζω ότι αν απαντήσουμε μία προς μία τις ερωτήσεις ε, που ο κύριος Ντεπρέ και ο κύριος Λεβαντόφσκι υποβάλλουν, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Τώρα βέβαια θα πρέπει να δούμε εν λεπτομερία το κείμενο, να δούμε το reflection paper, το working document. Ε, δεν είχαμε, ήταν πολλά τα έγγραφα, δεν μπορέσαμε να το δούμε ε, εν πλήρη λεπτομερία. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία τα οποία μου δίνουν τη δυνατότητα, την, την αίσθηση ότι θεωρούνται δεδομένα ε, και που δεν είναι πάντα έτσι. Το, αυτό το tax neutrality, η ουδετερότητα τι να σας πω, εμένα μου φαίνεται λίγο ε, σαν όνειρο αυτό, είναι λίγο χήμερα. Τι θα πούμε Εντάξει, λέμε ότι οπωσδήποτε η φορολογία δεν θα πρέπει να είναι επιθετική απέναντι στον πολίτη, οκ, αλλά ε, ουδετερότητα, ωραία, μιλάμε επίσης για ΦΠΑ, ε, μιλάμε για φόρο ε, στους, ε, στις μεταφορές ε, ή δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει tax neutrality ή πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο το λέμε γιατί ακούγεται ωραία, αλλά στην ουσία δεν είναι εύκολο. Άλλο θέμα τι θα κάνουμε με τους ίδιους πόρους. Δηλαδή θέλουμε ίδιους πόρους έτσι ώστε να μειώσουμε την εθνική συμβολή, γιατί στην προηγούμενη εντολή έγινε λόγος και γι' αυτό. Εγώ όμως έχω αμφιβολίες. Πρώτον το βλέπουμε και από την ορθή και από την ανάποδη ότι εάν ε, έχουμε κάποιες προτεραιότητες τι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, περισσότερα κονδύλια από όπου και αν έρθουν. Δεύτερον, ε, μπορεί να βρεθούμε σε μια δυσκολότερη κατάσταση, γιατί θα μειώσουμε τους εθνικούς ε, συμβιβασ... τους... την εθνική συνεισφορά και και ε, όμως ε, χρειαζόμαστε περισσότερους σπόρους. Επομένως ε, θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο. Δηλαδή ναι, να μειώσουμε ίσως τις συνεισφορές των κρατών μελών έτσι ώστε στη στιγμή της διαπραγμάτευσης να έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει και το είδαμε και στην ε, γεωργία, εξωτερική πολιτική, ανάπτυξη, επενδύσεις, ε, άμυνα, διαχείριση συνόρων, προσφυγική κρίση. Δεν έχουμε λεφτά. Άρα πρέπει να βρούμε χρήματα γι' αυτό. Ε, και μάλιστα έχουμε και πάμε το κεφάλι μας και το Brexit. Νομίζω ότι θα πρέπει να σπάσουμε κάποια ταμπού, πράγμα που δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τωμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές που ήταν πιο αποτελεσματικοί από μας. Έχετε ένα έγγραφο το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ και για τη μέθοδο που ακολουθήσατε γιατί αυτό το σύστημα των ερωτήσεων μπορεί να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε πολύ σωστά. Δεύτερη παρατήρηση. Θα κάνω την ίδια παρατήρηση ε, με την συνάδελφο. Δεν θα εκπλαγείτε. Εμένα με ενδιαφέρει η έννοια ε, και αναρωτιέμαι, προβληματίζομαι με την έννοια της ουδετερότητας. Ε, ουδετερότητα σημαίνει ότι δεν θα βαρύνουμε ακόμα περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν η απάντηση είναι ναι στο ερώτημα αυτό, τότε συμφωνούμε. Γιατί όντως και μέσω του ΦΠΑ και μέσω του της φορολογίας ε, εισοδήματος. Ε, οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι υπομένουν, ε, την υποστηρίζουν την, τη συμβολή. Εάν όμως ε, ουδετερότητα σημαίνει καθόλου επιπλέον φόροι και καθόλου επιπλέον πόροι, τότε δεν συμφωνούμε. Γιατί αν δεν έχουμε επιπλέον πόρους, τότε θα βρεθούμε στην κατάσταση που ανέφερε χθε ο Επίτροπος Έτιγκερ. Δηλαδή, ότι δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τον προπολογισμό που θέλουμε. Ε, το είχαμε αυτό και την προηγούμενη φορά και αναγκαστήκαμε να κάνουμε προσαρμογή ε, ε, πάνω σε προσαρμογή. Επομένως, ναι, ναι, έχουμε λιγότερα χρήματα από όσα θέλουμε, ε, ενώ ταυτόχρονα έχουμε περισσότερες ε, δαπάνες, ανάγκη δηλαδή για περισσότερες δαπάνες και έχουμε και τον Brexit. Και επομένως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να καθορίσουμε τα πλαίσια της νέας κατάστασης. Τρίτον, όσον αφορά την απανθρακοποίηση Το ανέφερε και ο Επίτροπος. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε προενεργητική στάση. Υπάρχουν πολλές ιδέες. Είναι αυτές του υψη, της ομάδας υψηλού επίπεδου υπό την προεδρία του κυρίου Μόντι. Υπάρχουν όμως και άλλες, ε, οι οποίες δεν ε, έγιναν δεκτές. Ε, είτε από την ομάδα, είτε έγιναν δεκτές από την ομάδα Μόντι, αλλά δεν έγιναν δεκτές από αλλού φορολογική ουδετερότητα για τους ε, ε, πολίτες δεν έχει καμία έννοια εάν δεν κάνουμε την προσαρμογή ε, του, του, άνθρακα στη, στα, σε σχέση με τα σύνορα. Γιατί διαφορετικά επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια έναντι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με την αποφυγή dumping, αλλά από την άλλη μεριά οι τρίτες χώρες ε, ε, πρέπει να πιστούν έτσι ώστε να κάνουν παραγωγές απανθρακωμένες όσο γίνεται περισσότερο, απανθρακοποιημένες. Και υπάρχει το ζήτημα των μεταφορών τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι αυτό το τα 0,1 cents ας πούμε ε, σε ένα αεροπορικό εισιτήριο ε, μπορεί να αποφέρει πάρα πολλά. και ακόμα και η αίσθηση που θα έχουν οι πολίτες απέναντι σε μια τέτοια ε, επιβάρυνση θα είναι πάρα πολύ λίγο. Un dollar, mais qui Quoi demander de mieux, on, de plus On demande plus à l'impôt et moins au compte. ένα, ε, ε, ένα πολύ μικρό ποσό ε, το οποίο όμως ούτε θα βαρύνει τους πολίτες και, ούτε θα, και τελικά θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Ε, όσον αφορά τώρα το ΑΕΠ. Euh, Εάν doit être évoquée. Όσον αφορά τώρα το, GNI, ΑΕ. Ε. δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε σημείο ανάπτυξης ε, που να μην χρειαζόμαστε ε, συσχέτιση με το ΑΕ. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να υπάρχει ελάφρυνση σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς ανάλογα κιόλας με το κράτος ε, για το οποίο ε, ε, μιλάμε. Όμως, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να προσθεθεί στο ερευνολογιό σας, αναρωτιέμαι εάν... αναρωτιέμαι περισσότερο για τον τρόπο υπολογισμού της συμβολής συνεισφοράς των κρατών μελών. Εγώ φοβάμαι ότι τα διορθωτικά στοιχεία στα οποία αναφέρεστε μπορεί να οδηγήσουν σε εκπτώσεις και περικοπές. Ίσως μπορούμε να αλλάξουμε την ερώτηση και να πούμε πώς θα υπολογίσουμε την συμβολή, τη συνεισφορά μονάχα επί τη βάση του ΑΕ ή σε αυτή τη βάση υπολογισμού θα προσθέσουμε και κάποια νέα στοιχεία αναφοράς ε, που θα συνδέονται ας με την εκπαίδευση, με το κλίμα, με το διοξείδιο του άνθρακος ε, που μπορεί να αποτελέσουν δείκτες ή σημεία αναφοράς, όπως θέλετε πέστε τα, θετικά, αντικειμενικά και που εν τέλει όλοι θα μπορέσουν να, ε, έχουν, να βγουν κερδισμένοι. αλλά κάπου ε, θα, πρέπει να, διασταυρωθούν αυτές οι δύο ε, τάσεις. Δηλαδή από τη μία λέμε ότι οι, οι των κρατών μελών θα μειωθούν, από την άλλη ότι τα έσοδα θα πρέπει να αυξηθούν. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτές οι δύο ε, γραμμές κάπου να τέμνονται δεν είναι δυνατόν αύριο να έχουμε ας πούμε 50% ίδιο πόρων ή 50% μείωση των εθνικών πόρων και 50% αύξηση των ιδίων πόρων. Ε, θα πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα ε, με, με σωστούς υπολογισμούς κλπ. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε ε, να δούμε, να θέσουμε το ερώτημα του τρόπου υπολογισμού της εθνικής συνεισφοράς. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές. Καλά το ξεκίνησε η κυρία Τομά. Έλεγε ότι εάν υπάρξουν φόροι ευρωπαϊκοί ας πούμε να μην αυξηθεί ταυτόχρονα ε, και το άχθος για τους πολίτες. Δηλαδή ναι ε, να υπάρχουν ενδεχομένως ευρωπαϊκοί φόροι αλλά ε, ο υπολογισμός να είναι τέτοιος ώστε να μειωθεί η εθνική συμβολή. Αυτό ε, κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να γίνει δημοφιλής ένας ευρωπαϊκός ε, πόρος ε, εάν του πούμε ότι θα πληρώνει τον ευρωπαϊκό φόρο και θα πληρώνει και τους φόρους. Ξέρω ότι εσείς θέλετε φόρους που να είναι άοσμοι και να, μην έχουν κανένα βάρος. Όχι, λέει η κυρία Τομάς. Θα απαντήσω. Σηκώσατε το γάντι της πρόκλησης. Θα είμαι σαφής όσον αφορά την, εταιρική φορολογία, corporate tax. Αυτό δεν σημαίνει επιπλέον προσπάθεια ε, ή φορό ε, για τους πολίτες, γιατί και η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση έχουν επιτρέψει ε, κάποιοι να μην πληρώσουν τα οφειλόμενα. Μιλάω για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες θα έπρεπε να πληρώσουν τουλάχιστον 12% γιατί αυτό νομίζω ότι είναι το πιο χαμηλό ποσοστό ε, του της εταιρικής φορολογίας στην Ιρλανδία ενώ στη Γαλλία είναι ας πούμε 33-35 σε άλλες χώρες. Επομένως οι μεγάλες εταιρείες θα έπρεπε να πληρώνουν ανάμεσα από 12 ή 33-35%. Όμως δεν πληρώνουν ε, απαραίτητα αυτό. Ξέρουμε ότι η Apple πληρώνει 0,00 κτλ. Επομένως δεν υπάρχει επιπλέον φόρος υπάρχει ή ε, μία διόρθωση έτσι ώστε να αποφύγουμε την, ε, τις εταιρείες οι οποίες φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν. Και δεν θα προσθεθεί λοιπόν αυτό πάνω σε κάποιον υφιστάμενο φόρο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παρουσιάσει κανείς τα πράγματα και πραγματικά πιστεύω ότι ναι, όντως αυτή είναι μια πραγματική συζήτηση, αλλά Ό,τι απόφαση και να πάρουμε δεν θα πρέπει να βαρύνουμε ε, τον φορολογούμενο πολίτη ε, ο οποίος ήδη πληρώνει αρκετά. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε οποιοδήποτε φόρο. Πρόεδρος, όσον αφορά τις πολυεθνικές, ορισμένες μεταξύ αυτών ε, δεν πληρώνουν όντως φόρο στην Ευρώπη, κάνουν φορολογικό ruling και αυτό φταίνε οι διοικήσεις, οι φορολογικές των ευρωπαϊκών χωρών. Η Google μέσω Ιρλανδίας και κάτω χωρών έχει μεταφέρει 4,5 δις της στις Βερμούδες. Αυτό έγινε γιατί οι Ευρωπαίοι ε, ε, είναι πάντα ε, εύκολοι και ευκολόπιστοι. Ας το πούμε έτσι. Και εδώ πραγματικά, πραγματικά θα πρέπει η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να ε, το μάθει και να μιλήσει. Ε, γιατί αν αφήσετε ας πούμε τον, ε, όπως κάνανε οι υπουργοί τον Ιούνιο του 2016 που συμμαζεύτηκαν εκεί για να συζητήσουν για το Λίξη και μετά έκαναν μια ανακοίνωση που έλεγαν ναι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φορά αποφυγή. Δηλαδή, δηλαδή μας φτύνουν στα μούτρα μας, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα εν πάση περιπτώσει, όντω είναι γεγονό ότι υπάρχει φορολογική ύλη η οποία εκφεύγει οποιασδήποτε φορολογική διοικήσεω και επομένω ε, δεν είναι δυνατόν αυτό να συνεχιστεί. Ε, ξέρουμε ότι όλη αυτή η φορολογική, η φορολογητέα ύλη η οποία δεν φορολογείται τελικά πηγαίνει και βρίσκει ένα ωραίο καταφύγιο στι βερμούδε. Παρακαλώ θα τελειώσω αυτό που έλεγε και θα σας δώσω το λόγο. Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει νομοθεσία η οποία ε, ε, ε, περιλαμβάνει μία ολόκληρη στρατιά ειδικών ρυθμίσεων, διατάξεων, υποδιατάξεων κτλ. Επομένως θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια στην, στα εθνικά φορολογικά συστήματα έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η σύγκληση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήθελα να σας, να σας διακόψω. Ναι, μας προκαλέσατε και απαντούμε στην πρόκληση αυτή. Υπάρχουν δύο ζητήματα είναι γεγονός ότι ε, ε, ε, οι φόροι που προτείνουμε τώρα είναι νέοι φόροι που θα αφορούν κάποιους τομείς που για την ώρα είτε δεν φορολογούνται αρκετά είτε φορολογούν, δεν φορολογούνται καθόλου. Δεν θα ψάξουμε τα λεφτά αυτά στις τσέπες άμεσα των φορολογούμενων αλλά τελικά λέει ο πρόεδρος αυτή στη δικιά τους, από τη δικιά του τσέπη θα βγούνε. Εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που Υπάρχει όμως και ένα πιο φιλοσοφικό ερώτημα, πιο βαθύ ερώτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι και να μην, φοβ... να μην ντρεπόμαστε για το ευρωπαϊκό ε, ε, σχέδιο. Εάν κάποια στιγμή ε, φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι για να χρηματοδοτήσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα πρέπει να φορολογήσουμε άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες, θα πρέπει να το πούμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν θέλουμε την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος και ε, ε, ονείρου, ε, να είμαστε έτοιμοι να φορολογήσουμε και να πληρώσουμε και φόρους αν πρέπει για την υγεία, για την ε, δημόσια ασφάλεια, για την πρόνοια να ε, πληρώσουμε κάποιους φόρους, ε, θα πρέπει να το κάνουμε. Γιατί τελικά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ανταποδίδει στον Ευρωπαίο πολίτη. Ναι, ξέρω ότι δεν πρέπει να κάνουμε άλματα. Πρώτα θα πρέπει να φορολογήσουμε ίσως τράπεζες. Είναι πιο εύκολο να πουλήσουμε μάλλον τη φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακα ή τη φορολόγηση των εκπομπών ή τη φορολόγηση των τραπεζών. Ακούγεται πιο ωραία χαϊδεύει πιο πολύ τα αυτιά, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σπάσουμε και αυγά. Πρόεδρος. Στις μεγάλες ε, δημοκρατίες ε, στην ουσία δημιουργήσαμε τα, τις εθνικές συνελεύσεις και τα κοινοβούλια έτσι ώστε να υπάρχει συνένεση όσον αφορά τα φορολογικά βάρη. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ντεπρέ. Σε σχέση με τα τελευταία που ακούστηκαν και σε σχέση με το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το ευρωπαϊκό ε, σχέδιο, και εγώ είμαι, ε, και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλήσουμε με καλά λόγια. Εγώ το κάνω και δεν διστάζω καθόλου. Ωστόσο, στο πρώτο σημείο ε, για το νομικό πλαίσιο, αναφέρεται ότι χρειάζεται η ομοφωνία του Συμβουλίου. Ομοφωνία του Συμβουλίου. Εντάξει, εγώ τώρα δεν πρόκειται να μιλήσω υπέρ μιας ε, ε, μηχανικής ε, διαφορετικής. Δεν θα ξεκινήσω τώρα μία διαδικασία για την οποία ξέρω ότι δεν πρόκειται να έχω ομοφωνία από το Συμβούλιο. Με αυτή την έννοια αναφέρουμε τη φορολογική ουδετερότητα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει επιπλέον ίδιος πόρος που θα βρεθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ε, επί της επικρατείας των κρατών μελών τότε η ε, συμβολή βάση του ΑΕΕ, του GNI θα πρέπει να μειωθεί. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μειωθεί η συμβολή κατα... σύμφωνα με το ΑΕ, γιατί διαφορετικά θα μας πούν, μας φορολογείται δύο φορές και δεν πρόκειται να το δεχτούν. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για ε, φορολογική ουδετερότητα. Δηλαδή όσο ανεβαίνει ο πρώτος πόρος, ε, θα κατεβαίνει ο, ε, ο, πόρος που σχετίζεται με το GNI, με το καθάριστο εγχώριο εισόδημα. Ε, και θα, δώσω, θα αφήσω τον Γιάννου να απαντήσει όπως θέλει σε αυτές τις άλλες ερωτήσεις. Πολύ σύντομα. Ε, να πω ότι ήδη έχετε αρχίσει να δίνετε απαντήσεις στα ερωτήματά μας, οπότε σας ευχαριστώ. σχέση, με το, σε σχέση με το ερωτηματολόγιο. Τώρα δεν θέλω να επιμείνω τη συζήτηση σε ό,τι αφορά την ε, φορά αποφυγή, αλλά ε, ούτως ή άλλως πάντοτε επανέρχεται αυτό το ζήτημα, όποτε τηθεί το ζήτημα της φοροαποφύγησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολογική ουδετερότητα, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη σχέση των ε, ιδίων πόρων ε, γενικότερα στο σύνολό τους και τη συνεισφοράς του καθάριστου εθνικού εισοδήματος. Ο πραγματικός στόχος εδώ είναι εξουδετερώσουμε αν θέλετε οποιασδήποτε κριτικές αντιδράσεις ε, απέναντι στην πρότασή μας. Ε, δηλαδή με βάση ε, το που κατέληξε η πρότασή μας το 2011 σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το στοιχείο της φορολογικής ουδετερότητας χωρίς επιπρόσθετα τέλη γιατί ούτως ή άλλως και αυτή η συνεισφορά του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος είναι οι συνεισφορές οι οποίες προέρχονται από φορολογικά έσοδα οπότε υπάρχει πάντοτε αυτή η σχέση. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρξει περαιτέρω ε, περιπλοκή αν θέλετε της φόρμουλας ε, υπολογισμού της συνεισφοράς χωρίς να υποτιμώ τα προβλήματα που υπάρχουν. Απλώς θα πρέπει να τηρήσουμε αυτή τη θέση γιατί με αυτόν τον τρόπο προωθούμε τη στάση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή η προσπάθεια που είχαμε κάνει για να υπάρξει άμεση σχέση μεταξύ του προϋπολογισμού και τη ε, συνεισφορά άμεσα από την πλευρά των ε, πολιτών, δυστυχώ δεν ανταποκρίνεται στο σημερινό επίπεδο εμπιστοσύνη των πολιτών μα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση. Αλλά ήδη με αυτόν τον τρόπο κάνουμε ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, θα ευχαριστήσω τους δύο Α, ο κύριο Ζάνη. Βάλει. Eh, Ζητώ συγγνώμη, δεν, ε, δεν ε, σύντομα, σύντομα παρακαλώ. Έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή. Πρέπει να προσπαθήσω να, ε, κατα... να, να δω πώς ε, ε, μπορούν ε, πραγματικά να γίνουν αποδεκτές από τις χώρες ε, οι ωραίες προτάσεις που έκανε η ομάδα του καθηγητού Μόντι. Το θέμα των, το, το θέμα των φόρων εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν με ομοφωνία και οι χώρες. Θα δούμε. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει παίξει στην ιστορία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Λείπει όμως κάτι από αυτήν την έκθεση. Λείπει μία ανάλυση της ε, κατάστασης στο εσωτερικό της Ευρωζώνης. Ε, θα με ενδιέφερε πάρα πολύ ε, κάτι τέτοιο γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να καταδειχθούν οι ανισορροπίες οι οποίες υπάρχουν. Να δούμε ότι υπάρχουν αυτές οι χώρες οι οποίες έχουν ας πούμε εμπορικό πλεόνασμα πάρα πολύ μεγάλο και που ίσως αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο στο προϋπολογισμό είτε της Ευρωζώνης είτε του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να υπενθυμίσουμε επίσης ε, ότι ε, αυτές οι οικονομικές ανισορροπίες είναι ακριβώς το στοιχείο το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτάσεις ε, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ενδιαφέρουσες, Αυτές, ας πούμε για τον φόρο του διοξιδίου του άνθρακος. Βλέπω ιδιαίτερα μη δημοφιλή μια φορολόγηση επί των ε, των ε, ορυκτών καυσίμων. Κοιτάξτε, εγώ έχω καθαρά ε, συμβαστική και τάση και τάση συνεργασίας και το λέω σαφώς και στον συνάδελφο Ντεπρέ. Ε, και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό μου φαίνεται λίγο ε, χειμερικός αυτός ο προϋπολογισμός. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτού του είδους την πρόταση φορολόγησης οι πολίτες να την εννοήσουν, να την εκλάβουν ως επιπλέον φορολόγηση. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στους ε, πολίτες ε, ε, τι σημαίνει ακριβώς αυτή η αύξηση, γιατί θα είναι νομίζω πάρα πολύ επικίνδυνο να θεωρήσουν ότι θα αυξηθούν οι φόροι και επομένως θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η οικονομία η οποία χυμάζει για την ώρα και η οποία τώρα σιγά σιγά παίρνει λίγο τα πάνω της. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Βλέπω ότι συγκλίνουν οι απόψει, βεβαίω το κυρίαρχο ερώτημα είναι τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Ποια Ευρώπη θέλουμε να δώσουμε στους ε, πολίτες ε, μας. Με ποιο τρόπο θέλουμε να απαντήσουμε στις απαιτήσεις τους, στις ιδέες τους. Αν θέλουμε αυτήν την ε, δυνατή Ευρώπη, η οποία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, θα πρέπει να οικοδομήσουμε και έναν σωστό προϋπολογισμό ε, με τα απαραίτητα έσοδα. Η φορολόγηση και οι φόροι συζητιούνται σε μια δημοκρατία και δεν θα πρέπει βεβαίως να πέσουμε στην παγίδα να, μιλάμε, να σκεφτόμαστε περισσότερο τους φόρους και λιγότερο τους φορολογούμενους. Δύο λόγια να πω, κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Δεπρέ δεν είναι μόνο οι φόροι, υπάρχουν και έσοδα. Μία συμβουλή στην Κομισιόν. δυόμιση δις, ε, εκατομμύρια να επιβάλλει πρόστιμο σε μία πολυεθνική, στην ουσία ε, βγάζει τα λεφτά του Brexit. Πριν φύγετε συνάδελφοι να σας πω ότι έχουμε δύο ανθρώπους ε, εν συγκινήσει. Η Φάμπια Τζόνς ε, ανέλαβε την ε, δίκη, την, έγινε επικεφαλής στην γραμματεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών τον Ιανουάριο του 2015. Για δυόμιση χρόνια λοιπόν με μεγάλη αποτελεσματικότητα, διακριτικότητα, ε, πάντα ε, ε, με χαμόγελο, το οποίο έκρυβε όμως την πυγμή της και τον δυνατό της χαρακτήρα, λειτουργήσε εδώ στην Επιτροπή. Τώρα θα πάει σε μια άλλη υπηρεσία ως εμπειρογνώμων και θα ήθελε λοιπόν με την ευκαιρία της εξόδου της, της αναχώρησής της, να της ευχηθώ τα καλύτερα. Να την ευχαριστήσω και να σας πω ότι αυτή ε, η σιδερένια πυγμή στο βελούδινο γάντι της μας ήταν πάντα ε, ιδιαίτερος ε, ευχάριστη. Τη θέση της αναλαμβάνει μια άλλη συνάδελφος, τη, τη Φάμπια, την οποία να καλωσορίζουμε. Ευελπιστούμε ότι θα είναι καλά στην καινούργια θέση. Ε, και να πούμε ότι η Φάμπια είναι η πιο Βελγίδα, ε, η πιο Βελγίδα Βρετανίδα. Και εξ ονόματός σας θα την φιλήσω στα βρωτά. Επόμενη συνεδρίαση 10 και 11 Ιουλίου. Ε, αυτά λοιπόν.